Let us start with our normal meeting. The first point... Ας αρχίσουμε λοιπόν με την συνεδρίαση μας. Είχαμε την συνεδρίαση των συντονιστών. During, during uh, the time, you will get via email. Πρέπει να σας πω ότι θα σας στείλω με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο τα αποτελέσματα της συνεδρίασης των uh, συντονιστών. Ε, άμα θέλετε μπορούμε και να τα τυπώστε τα μάλλον εσείς, διαβάστε τα και να ξέρετε ότι πρέπει έτσι κι αλλιώ να εγκρίνουμε αυτές τις αποφάσεις μέχρι το τέλος της συνεδρίασης. Οπότε μελετήστε τα και πείτε μου αν έχετε αντιρρήσεις. Σημείο 2, είπαμε έγκριση της ημερήσιας διάταξης, συμφωνείτε εντάξει, σημείο 3, έγκριση των πρακτικών της συνεδρίας στις 5 και 6 Οκτωβρίου, αν μέχρι το τέλος της συνεδριάσεως δεν ε, έχετε αντιρρήσεις, θεωρούνται εγκεκριμένα. Και έτσι συνεχίζουμε. Αλλά θέλω προηγουμένως να σας υπενθυμίσω... Α, μια στιγμή, μια στιγμή, γερμανικά συνεχίζει η Πρόεδρος. Είχαμε λοιπόν τη συνεδρία συντονιστών που η Πρόεδρος και θα σας διαβιβάσω τα συμπεράσματα με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο το μεσημέρι για να μπορέσετε να σχολιάσετε ή τυχόν υποβάλλατε ε, τροπολογίες ή σχόλια και παρατηρήσεις. Ε, ζητήσαμε από την Κομισιόν να συντάξει μία μελέτη για την ε, πολιτιστική πολυμορφία στο μουσικό τομέα. Και αυτή η μελέτη λοιπόν έχει ολοκληρωθεί και θα συζητηθεί σήμερα στα πλαίσια της νομικής... Α, στις 2 Δεκεμβρίου, στις 2 Δεκεμβρίου, όχι σήμερα. Τετάρτη Στι 3 διορθώνει η κυρία Πακ. Τετάρτη στι 2 Δεκεμβρίου στι 3 η ώρα το απόγευμα. Τετάρτη 2 Δεκεμβρίου 3 η ώρα νομική επιτροπή. Το θέμα είναι collective societies και μουσική επικοινομορφία. Ε, χαίρομαι σήμερα που μπορούμε σήμερα να καλωσορίσουμε τον ε, νέο επίτροπο μετά τις 19 ε, Σεπτεμβρίου, ο κύριος Σεύκοβιτς, ε, ο νέος επίτροπος είναι μαζί μας σήμερα, ο οποίος είχε στο παρελθόν μια λαμπρή διπλωματική καριέρα, η οποία του επέτρεψε να ασχοληθεί με πολλά κοινοτικά θέματα και μάλιστα σε έναν τομέα, ο οποίος έχει άμεση σχέση με τις, τους ανθρώπινους πόρους και τις ανθρώπινες επαφές. Εν συνεχεία ανακατεύθηκε στην πολιτική της ε, χώρας του και τώρα τον, από τον Οκτώβριο, τέλη Σεπτεμβρίου, αρχές Οκτωβρίου και πέρα είναι ένας από τους επιτρόπους μας. Αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε σε μια δύσκολη εποχή ορισμού επιτρόπων και έχουμε διαλέξει μια πάρα πολύ ρεαλιστική οδό. Είπαμε θα περιμένουμε μέχρι ότι ε, έχουν ονομαστεί όλοι οι επίτροποι και μετά θα γίνουν οι ακρόασει. Δεν θα κάνουμε σήμερα ακρόαση ε, στον κύριο Επίτροπο, ο οποίο μπορεί σε δύο εβδομάδε να μην είναι πια Επίτροπος. Ε, ούτε εμεί το ξέρουμε βέβαια αν θα είναι ή δεν θα είναι, άρα λοιπόν δεν θέλουμε να, να κάνουμε την ακρόαση σήμερα, Απλώ θα μιλήσουμε σήμερα μαζί του, θα κάνουμε ένα διάλογο. Έχει ήδη την εμπειρία μια εισαγωγή ε, αυτή τη ε, θέση, είναι εμπειρογνώμο στον τομέα του και θα έχουμε ασφαλώ την ευκαιρία να συζητήσουμε μαζί του. Χαίρομαι επίση που είναι μαζί μα κυρία Κεντά. Πού είναι, την είδα προηγουμένω. ωραία. Είναι εδώ η Γενική Διευθύντρια κύριος Τίσον, ο Νόρβερ Σούμπερ και ο κύριος Πάβελ Κόσεκ. Είναι εδώ λοιπόν όλες μας οι εξέχουσες προσωπικότητες και τώρα θέλω να δώσω το λόγο στον Επίτροπο κύριο Σεύκοβιτς να μας μιλήσει για την εμπειρία του του τελευταίου μηνός και να μας παρουσιάσει ορισμένα σχόλια από πλευράς Κομισιόν. Θα είμαστε είναι ευπρόσδεκτος και αναμένουμε με ανυπομονησία τα σχόλιά του. Θα έχετε την υποστήριξή μας να είστε βέβαιος προς ε, οπουδήποτε μετακινηθείτε ή όχι. Ε, και έχουμε απόλυτη εμπιστοσύνη σε εσά. Παρακαλώ, έχετε το λόγο. Σα ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε. Som naozaj e, veľmi rád za toto veľmi vrele e, v Európskom e, parlamente a chcem sa poďakovať za možnosť stretnutí s πάρα πολύ που βρίσκουμε σας στο νέο κοινοβούλιο και θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για τη συνεργασία στον τελευταίο μήνα. Οι συνεδριάσεις με ενέπνευσαν, ήταν πάρα πολύ δημιουργικές και ευχαριστώ ιδιαίτερα τη Γενική Διευθύντρια κυρία Καντάν, η οποία ήταν πραγματικά, με υποστήριξε έντονα, με βοήθησε πάρα πολύ ε, κατά τη διάρκεια των συναντήσεων μου και το, ε, στα meetings που είχα στο, στη καινούργια μου θέση. Σας ευχαριστώ πολύ και για την υποδοχή που μου επιφυλάξατε εδώ πέρα και για τα καλά λόγια της Προέδρου. Χάρη σε διάφορες επαφές που είχα μαζί σας όλο αυτό το καιρό, να ξέρετε ότι Κατάφερα να προχωρήσω πολύ με το χαρτοφυλάκιο μου αυτό για την εκπαίδευση, την νεότητα, τον αθλητισμό, την κατάρτιση. Έχει τεράστιο δυναμικό το χαρτοφυλάκιο αυτό για το μέλλον. Και μπόρεσα να δουλέψω πάρα πολύ ακριβώς επειδή είχα καλή συνεργασία με το Κοινοβούλιο. Ξέρω ότι πολλά από τα προγράμματα που προωθήσαμε δεν θα τα είχαμε προωθήσει με τον ίδιο τρόπο αν δεν είχαμε τη δικιά σας τη στήριξη, αν δεν είχαμε τις δικές σας τις προτάσεις και δεν θα μπορούσαμε να είχαμε κάνει τόσο όσα κάναμε σε ευρωπαϊκό επίπεδο χωρίς τη στήριξη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ε, κατά τη διάρκεια των δύσκολων δημοσιονομικών συζητήσεων που λαμβάνουν χώρα ετησίως. Τα τελευταία πέντε χρόνια, ειλικρινά, καταφέραμε πολλά. Και αν έπρεπε να συνοψίσω τα κύρια επιτεύγματα των τελευταίων πέντε ετών, θα έλεγα ότι κανείς δεν αναρωτιέται πια αν μπορεί να φέρει προστιθέμενη αξία στον τομέα της εκπαίδευσης και της κατάρτισης η Ευρωπαϊκή Ένωση. Και αυτό γιατί είναι πια σαφές ότι η Ευρώπη μπορεί να κάνει πολλά. Αυτό έχει αποδειχτεί ξανά και ξανά παρά την πρόσφατη κρίση. Ας δούμε λοιπόν Ποιοι είναι οι στόχοι μας, τα προγράμματά μας στον τομέα του πολιτισμού και της εκπαίδευσης. Κάθε χρόνο πάνω από 500.000 ε, Ευρωπαίοι πολίτες ε, εποφελούνται από τα προγράμματά μας ε, αυτά και από τα κονδύλια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι πάνω από 1% προπολογισμό που πάει εκεί από το συνολικό ευρωπαϊκό προπολογισμό. Πάντα με τη βοήθεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ελπίζουμε να καταφέρουμε στο μέλλον το ποσοστό αυτό να αυξηθεί. Η στρατηγική της Λισαβόνας τώρα δείχνει με σαφήνεια ότι θέλουμε να έχουμε μια ανταγωνιστική οικονομία στην Ευρωπαϊκή Ένωση που να είναι προς όφελος ε, του κόσμου, της ε, εκπαίδευσης, της κατάρτισης και του πολιτισμού. Αυτά φαίνονται και από τα επίσημα έγγραφα τα οποία ε, εκδίδουμε. Έχουν γίνει πολλές σοβαρές συζητήσεις για όλα αυτά, τα οποία οδήγησαν στα συμπεράσματα του Συμβουλίου που έχουμε ήδη από το 2005. Κάτι άλλο πάρα πολύ σημαντικό θα ολοκληρωθεί μέχρι τα τέλη της χρονιάς. Δηλαδή όλες αυτές οι τεράστιες προσπάθειες που έχουν γίνει στο, για το Ευρωπαϊκό ε, Τεχνολογικό Ινστιτούτο θα υλοποιηθούν πια με την πρώτη επιλογή που θα γίνει των ε, κοινοτήτων αυτών καινοτομία και τεχνολογίας. Είναι η εφαρμογή του τριγώνου της γνώσης, δηλαδή η έρευνα, η γνώση και η καινοτομία. Όταν κοίταζα τα στοιχεία, τι έχουμε πετύχει δηλαδή τα τελευταία χρόνια, με εξέπληξε το εξή. Το 87 μόνο 3.000 ε, προγράμματα έρασμος έχουμε. Μπορεί αυτό το νούμερο να συγκριθεί με τις 160.000, όχι βέβαια, αλλά εκείνη την εποχή κανένας δεν μπορούσε να φανταστεί πόσο μεγάλη επιτυχία θα είχε το πρόγραμμα Έρασμος μέσα σε 20 χρόνια. Να όμως, οι φιλοδοξίες μας Πέτυχαν και γίνονται μεγαλύτερες ε, όσο περνάει ο καιρός. Επίσης, πάρα πολύ καλή συνεργασία είχαμε και με τα κράτη-μέλη και ιδιαίτερα για τα προγράμματα προσχολικής ηλικίας. Όντως, μας ε, ζητιέται όλο και περισσότερο να φροντίζουμε για τα παιδιά σε προσχολική ηλικία, γιατί παίρνουν έτσι καλές συνήθειες, πώς να μάθουν να μαθαίνουν, Όλα αυτά αποδεικνύονται από τις μελέτες που έχουν γίνει μέχρι τώρα και αυτό βέβαια βοηθάει και την απασχόληση. Αυτά είναι επιτεύγματα, χωρίς όμως να σημαίνει ότι δεν έχουμε πολλές προκλήσεις μπροστά μας. Και αυτό πρέπει να το καταλάβουμε καλά. Έχουμε την μελέτη PISA που μας βοηθάει να δούμε πιο ξεκάθαρα τις προκλήσεις που έχουμε. Πρόκειται για τον αναλφαβητισμό. Τα πράγματα πρέπει να βελτιωθούν στον τομέα αυτό. Είναι κρίμα που δεν μπορούμε να πετύχουμε τους στόχους μας ε, ήδη από τα πρώτα χρόνια του σχολείου. Ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι εμείς θέλουμε μέχρι το 2010 να πετύχουμε το στόχο μας. Θα δούμε. Ελπίζω ότι η νέα Επιτροπή θα μπορέσει να πετύχει το στόχο. Τώρα, ποια είναι η μεγάλη πρόκληση που βλέπω εγώ για το μέλλον αυτή είναι πώς θα βελτιωθεί η ποιότητα του εργατικού μας δυναμικού. Και αυτό γιατί σήμερα έχουμε πάνω από 80 εκατομμύρια Ευρωπαίους πολίτες οι οποίοι έχουν χαμηλά προσόντα. Πρόκειται για το 1 τρίτο του εργατικού δυναμικού στην Ευρώπη. Δεν είναι δυνατόν να συνεχίσουμε έτσι στο μέλλον. Είναι ξεκάθαρο ότι μια οικονομία που βασίζεται στη γνώση πρέπει να επιταχύνει τους ρυθμούς της και ότι οι άνθρωποι αυτοί μέσα σε μια τέτοια οικονομία της γνώσης θα βρεθούν στο περιθώριο όλο και περισσότερο. Τι πρέπει λοιπόν να κάνουμε. Πρέπει να δουλέψουμε παράλληλα. Δηλαδή από τη μια να βελτιώσουμε τη διδακτική ύλη στα σχολεία, ώστε να είναι περισσότερο στοχευμένη προς την ε, αγορά και την οικονομία και από την άλλη μεριά πρέπει να κάνουμε περισσότερες προσπάθειες όσον αφορά τη διαβίου κατάρτιση ή την εκπαίδευση των ενηλίκων, ώστε να μπορέσουν να αποκτήσουν νέα προσόντα και έτσι να έχουν στη διάθεσή τους νέες ευκαιρίες για να ε, απασχοληθούν και να μην μείνουν στην ανεργία. Είχαμε πρόσφατα και την οικονομική κρίση. Όλοι περίμεναν ότι μόνο οι οικονομικές υπηρεσίες θα πληγούν. Η αλήθεια όμως είναι ότι οι άνθρωποι με χαμηλά προσόντα και οι νέοι είναι εκείνοι οι πλήττονται περισσότερο από την οικονομική κρίση. Άρα πρέπει να τους βοηθήσουμε. Πρέπει να βρούμε συνταγές για να ξεπεράσουμε αυτή τη δυσκολία. Θετικά επίσης μπορούμε να αξιολογήσουμε και τις αντιδράσεις των κρατών ε, μελών στην πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ώστε να συμπεριληφθεί στην ε, διδακτέα ύλη κάτι που έχει να κάνει με νέες θέσεις απασχόλησης, νέα επαγγέλματα, νέες ιδέες, καινοτομία. Πρέπει δηλαδή τη μέθοδο εκμάθησης στα σχολεία και την ύλη που διδάσκονται τα παιδιά στο σχολείο να την προσαρμόσουμε στις πραγματικές ανάγκες μιας πραγματικής αγοράς εργασίας. Πήγα στο Πανεπιστήμιο του Λούντ στη Σουηδία πρόσφατα και πραγματικά ήταν μεγάλο προνόμιο για μένα να δω εκεί τους ε, φοιτητές ε, του προγράμματος Έρασμος. Ε, και είδα πόσα πολλά προσφέρει το πρόγραμμα αυτό στους νέους. Πρώτα απ' όλα μαθαίνουν καλύτερα ξένες γλώσσες. Έπειτα γυρνάνε πίσω στις χώρες τους με περισσότερη εμπιστοσύνη στον εαυτό τους έχουν ε, μια πιο θετική και καλύτερη προσέγγιση στην ε, ζωή μέσα στην κοινωνία. Αυτό είναι κάτι που πρέπει να το στηρίξουμε και να κάνουμε ακόμα περισσότερο. Γι' αυτό χάρηκα πάρα πολύ που είδα ότι και ο πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής εξέφρασε τις σκέψεις του για αυτή τη θετική εμπειρία στις κατευθυντήριες γραμμές της Επιτροπής και πήρε την πρωτοβουλία για το πρόγραμμα Youth on the Move, η νεολαία εν κινήσει. Δηλαδή να μπορούν έτσι φοιτητέ να ε, περνάνε κάποιο κομμάτι το σπουδό του στο εξωτερικό, με περισσότερη κινητοποίηση πόρων από την Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά και από τα κράτη-μέλη, αλλά και από το περιφερειακό επίπεδο. Και πρέπει να συμμετέχει και ο ιδιωτικό τομέα σε αυτό, γιατί όχι. Όπω επίση και παιδαγωγικά Ινστιτούτα. Με αυτή την κινητικότητα όμω θέλουμε και περισσότερη κινητοποίηση. Δηλαδή οι νέοι να είναι πιο δραστήριοι μέσα στους δημοκρατικούς θεσμούς. Πώς δηλαδή ε, διαχειριζόμαστε τα σχολεία, να συμμετέχουν στην πολιτική ζωή των χωρών τους. Είδα χτες τα ντόμινο που πέφτανε στο Βερολίνο, τα κομμάτια αυτά. Και είδα ότι 20 χρόνια πέρασαν όντω από τότε που έπεσε το τείχος του Βερολίνου και διαπιστώνω ότι για πρώτη φορά έχουμε μια νέα γενιά στην Ευρώπη η οποία γεννήθηκε μέσα σε μια ενωπημένη Ευρώπη. Δηλαδή που δεν ζήσαν, δεν γνωρίσανε την εποχή εκείνη που ήταν μοιρασμένη η Ευρώπη, που υπήρχαν έλεγχοι, που υπήρχαν τείχοι. Όλα αυτά έκαναν ε, τους νέους εκείνη την εποχή να μην γνωρίζουν τι συμβαίνει από την άλλη μεριά. Δεν υπάρχει πια αυτό έχουμε την πρώτη πραγματικά ευρωπαϊκή γενιά η οποία μπορεί να συμμετέχει περισσότερο στην ευρωπαϊκή ζωή. Έτσι πρέπει να φτιάξουμε τις προϋποθέσεις για να τη βοηθήσουμε να συμμετέχει στην ευρωπαϊκή ζωή. Επίσης είμαι ιδιαίτερα ικανοποιημένος για την πρόοδο που πετύχαμε τα τελευταία χρόνια στον τομέα του πολιτισμού. Χάρη και στο έτος της δημιουργικότητας και καινοτομίας δείξαμε τι δυνατότητες έχουμε για τη δημιουργία και για επιχειρήσεις που έχουν να κάνουν με τη δημιουργία. Ο πολιτισμός είναι ένα φαινόμενο που πρώτα απ' όλα ενώνει την Ευρώπη, τις ευρωπαϊκές χώρες, τα ευρωπαϊκά έθνη. Είναι επίσης κάτι σαν πρέσβυρα ο πολιτισμός της Ευρώπης προς τα υπόλοιπα μέρη του κόσμου. Αλλά αυτό έχει και οικονομικά ωφέλη. Από πρόσφατες μελέτες βλέπουμε ότι ο πολιτισμός και οι επιχειρήσεις που έχουν να κάνουν με τη δημιουργία συνεισφέρουν στο τζίρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο Ευρωπαϊκό ΕΠ, πάνω από 1,6%. Το οποίο στο 100% είναι παραπάνω από ότι μας αποφέρουν τα αλκοολούχα ποτά ή τα τσιγάρα. Άρα υπάρχουν τεράστιες δυνατότητες σε αυτό το τομέα. Πρέπει να συνεχίσουμε να δουλεύουμε συνεπώς ώστε οι προϋποθέσεις να είναι καλύτερες, πιο ξεκάθαρες και να δείξουμε το δρόμο πώς θα αντιμετωπίσουμε και το θέμα της ε, πνευματικής ιδιοκτησίας και της καταχρήσης που γίνονται σε αυτό. Για να μείβονται καλά οι καλλιτέχνες, οι συγγραφείς και να διασφαλίσουμε όσο γίνεται περισσότερο συγχρόνως πρόσβαση των Ευρωπαίων πολιτών στον πολιτισμό και στη γνώση. Πρέπει να βρούμε έναν ευρωπαϊκό τρόπο, γιατί δεν μπορούμε να βασιζόμαστε στις αποφάσεις των Αμερικανικών δικαστηρίων, αυτή θα είναι μια από τι προτεραιότητε της επόμενη Ευρωπαϊκή Επιτροπή, πιστεύω. Αυτό βέβαια καταδεικνύεται ακόμα περισσότερο και από την πρόσφατη συζήτηση που έχει γίνει για το Google και για τι δικαστικέ υποθέσει που εκκρεμούν ακόμα στα Αμερικανικά δικαστήρια. Σίγουρα και αυτό θα βρεθεί ε, στο τραπέζι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής μέσα στους επόμενους μήνες. Θέλω να σας ευχαριστήσω επίσης όλους για την πρωτοβουλία που πήρατε όσον αφορά την Ευρωπαϊκή Κληρονομιά. Γιατί και αυτή είναι μια πρωτοβουλία που μπορεί να βοηθήσει. Έρχεται από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και μπορεί πραγματικά να βοηθήσει διακυβερνητικές ε, διαδικασίες για αυτό το πραγματικά ευρωπαϊκό εγχείρημα. Το σήμα αυτό της Ευρωπαϊκής Κληρονομιάς θα συμπληρωθεί και έτσι θα μπορέσουν διάφοροι χώρες στην Ευρώπη να αποκτήσουν αυτό το σήμα. Και έτσι θα μπορούμε να φτιάξουμε και κάποια μικρά πακετάκια με πληροφορίες για να ενημερωθούν οι πολίτες, να ξέρουν ο κάθε αρχαιολογικός χώρος ή ο κάθε πολιτιστικός χώρος τι ακριβώς είναι. Αυτό βοηθάει και την εκπαίδευση αλλά και τοπικά τις διάφορες περιφέρειες να κερδίσουν και περισσότερα χρήματα. Θέλω να ευχαριστήσω τον κύριο Σκούρη επίσης για την δικιά του επικοδομητική προσέγγιση και για τις ιδέες του προκειμένου να συμπληρωθεί το έργο μας για την προετοιμασία του Ευρωπαϊκού Έτους Εθελοντισμού. Όσοι ξέρουν από πού έρχεται και τι έχει κάνει στη ζωή του θα εντυπωσιαστεί από την μεγάλη του εμπειρία, από τις δραστηριότητές του στον τομέα του εθελοντισμού. Ξέρω ότι το θέμα αυτό βρίσκεται λοιπόν σε καλά χέρια και περιμένουμε να ετοιμαστεί η προπαρασκευαστική δουλειά για να προχωρήσουμε στην ομοθεσία στο Συμβούλιο. Τώρα έρχομαι στον αθλητισμό. Με τον αθλητισμό υπάρχουν πολλές προσδοκίες. Και χαιρόμαστε πολύ στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή που έχουμε αυτή τη νέα αρμοδιότητα. Θέλουμε να χτίσουμε πάνω στην Λευκή Βίβλο μας και να έχουμε διαβουλεύσεις με όλους τους εμπλεκόμενους, ώστε να καταλήξουμε σε νέα ανακοίνωση για τον αθλητισμό του χρόνου. Θέλουμε να χρησιμοποιήσουμε όσο γίνεται περισσότερο τις δυνατότητες που έχουμε για αυτή τη νέα αρμοδιότητα. Με το πόσο σημασία έχει για την υγεία, για παράδειγμα, αθλητισμός για τα παιδιά. Και συγχρόνως θέλουμε να δημιουργήσουμε ένα υγιές νομοθετικό πλαίσιο για τις αθλητικές δραστηριότητες. Θέλουμε ε, να σεβόμαστε την ιδιαιτερότητα του αθλητισμού, την αυτονομία των ε, αθλητικών συλλόγων και συγχρόνως η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να διασφαλίσει και την τήρηση του νόμου αλλά και τα δικαιώματα των Ευρωπαίων πολιτών. Κύριε Πρόεδρε, αυτή νομίζω ότι θα είναι μια από τις κύριες προτεραιότητές μας και σίγουρα προτεραιότητα θα είναι στην επόμενη Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Θέλω να ολοκληρώσω με το τι θα κάνουμε στο μέλλον. Θέλουμε να στηρίξουμε τα κράτη-μέλη. Θέλουμε να τα βοηθήσουμε να εξυγχρονίσουν την σχολική εκπαίδευση, να στηρίξουμε τους καθηγητές και την διαβίου κατάρτιση. Θέλουμε επίσης να προωθήσουμε και να στηρίξουμε την κινητικότητα. Αλλά θέλουμε και κινητοποίηση των νέων. Θέλουμε επίσης να στηρίξουμε τις ε, πολιτιστικές επιχειρήσεις, κάθε επιχείρηση η οποία ασχολείται με τη δημιουργία. Θέλουμε να στηρίξουμε τους συγγραφείς, τους καλλιτέχνες και να φροντίσουμε να υπάρχει μεγάλη πρόσβαση του κοινού στα πολιτιστικά αγαθά. Επίσης, να ολοκληρώσουμε το έργο μας για το σήμα της πολιτιστικής κληρονομιάς. Και όπως είπα και πριν από λίγο, θα κάνουμε ό,τι μπορούμε για να χρησιμοποιήσουμε τις νέες αυτές αρμοδιότητες που έχει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στον τομέα του αθλητισμού όσο γίνεται περισσότερο. Κύριε Πρόεδρε, σας ευχαριστώ πολύ και θα ακούσω τώρα τα δικά σας σχόλια και τις ερωτήσεις σας. Είμαι έτοιμος ό,τι θέλετε να σας απαντήσω. Ευχαριστώ κύριε Επίτροπε. Έχουμε 30 λεπτά στη διάθεσή μας. Δεν θέλω να πω εγώ τίποτα, για να μην σας ε, καθυστερώ. Η κυρία Τρίπελ, πρώτα, ο κύριος Φίσας, η κυρία... Δεν μπορούμε να διαβάσουμε. Η κυρία με το κόκκινο, η κυρία στο μέσον, η κυρία Μπαντιά και συνεχίζουμε. Τηλεγραφικά παρακαλώ. Η κυρία Τρίπελ. Σε ευχαριστώ, Ντόρις. Σας ευχαριστώ κύριε Επίτροπε Σεύκοβιτς για την πολύ επικοδομητική σας παρέμβαση η οποία περιείχε πάρα πολλά θετικά στοιχεία. Θα ήθελα να, να, πω μόνο ότι είμαι πάρα πολύ ευτυχής με αυτό που είπατε για, την ε, πνευματική, για, την, ε, για το copyright και ότι θα πρέπει να εργαστούμε στο να, για να δημιουργήσουμε ένα, ε, μια ευρωπαϊκή άδεια ευρεσιτεχνίας και επίσης ε, χαίρομαι ιδιαίτερα που αναφέρετε τη νέα γενιά και την υποστήριξη που πρέπει να τους δώσουμε ιδιαίτερα για να συμμετωθούν στο βιομηχανικό τομέα, στον οικονομικό τομέα. Όλα αυτά τα οποία αναφέρετε βεβαίως καλύπτονται από την αναθεώρηση του προϋπολογισμού. Εάν θέλουμε να επενδύσουμε περισσότερες πιστώσεις στην ε, διαρκή ε, εκπαίδευση, στα προγράμματα Εράσμους και στη νέα γενιά, τότε θα πρέπει το Σώμα των Επιτρόπων να ασκήσει πίεση ώστε να έχει μια πολιτική επίδραση στην όλη διαδικασία αναθεώρησης του προϋπολογισμού διότι από εκεί εξαρτάται. Πρέπει λοιπόν να φροντίσουμε να ασκήσουμε τη σχετική πίεση μέσω των επιτρόπων στον προπολογισμό και την αναθεώρηση για να μπορέσουμε να επιτύχουμε αυτή, αυτά τα κονδύλια, να εξασφαλίσουμε αυτέ τι πιστώσει. Θα πρέπει λοιπόν εσεί ω Επίτροπο να φροντίσετε να προβάλλετε περισσότερο αυτού του τομεί τη πολιτική μα και ειδικά τώρα στα πλαίσια τη στρατηγική τη Λισαβόνα πρέπει οπωσδήποτε να διαθέσουμε περισσότερα χρήματα για αυτούς τους τομείς μέσα στα πλαίσια Λισαβόνας. Η πρόεδρος. Ε, ο κύριος Φίσας. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ πολύ κύριε Επίτροπε που είσαστε εδώ. Θα είμαι σύντομος. Συμφωνώ πολύ με τον Επίτροπο, με τόσα είπε, αλλά θέλω να αναφερθώ σε ένα σημαντικό για μένα θέμα. Πρόκειται για τη, τους μεκίνες, για το sponsoring, για τις επιχειρήσεις και όχι μόνο που μπορούν να στηρίξουν τον αθλητισμό ή την εκπαίδευση. Θέλω λοιπόν μέσω του συντονιστή μας του κύριου Σκούρη να ζητήσουμε από τις υπηρεσίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου να μας ετοιμάσουν μια μικρή εκθεσούλα γι' αυτό και να έχουμε κάποια σύγκριση. Τι γίνεται στις ΗΠΑ με τη Μεκίνη, τι γίνεται στην Ευρώπη. Διότι τα χρήματα δεν είναι πολλά, πιστεύω. Και θα ήταν σημαντικό να μπορέσουμε να αναλάβουμε κάποια πρωτοβουλία προς αυτή την κατεύθυνση, δηλαδή να ζητήσουμε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να το κάνει. Έρχομαι τώρα στον αθλητισμό. Προσωπικά έχω μια εμπειρία γιατί στη Μαδρίτη οργάνωσα κάποιο αθλητικό γεγονός για μαθητές. Και ήταν πραγματικά πάρα πολύ καλό όσον αφορά την ένταξη των μεταναστών, γιατί αποδείχτηκαν πρωταγωνιστές τελικά στις ομάδες τους. Δεν ξέρω αν είναι περίπλοκο ή όχι, αλλά δεν θα μπορούσαμε να κάνουμε κάτι αντίστοιχο σε ευρωπαϊκό επίπεδο, δηλαδή κάποιους ε, αγώνες ε, πανευρωπαϊκούς με παιδιά σε σχολική ηλικία. Dzień e, Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ. Ε, είναι πάρα πολύ ενδιαφέροντα όλα αυτά που μας είπατε. Ε, αυτό που θα ήθελα να μάθω από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι ε, τι σκοπεύει να κάνει και με τις ε, χώρες που βρίσκονται στα ανατολικά της Ευρώπης. Μιλήσατε βεβαίως αγγλικά και οι περισσότεροι μεταξύ ημών μιλά, μιλούμε την ωραία γλώσσα του Σέξπιρ, αλλά νομίζω ότι καλό θα ήταν να χρησιμοποιήσετε και την δική σας γλώσσα, γιατί αυτού του είδους η Ευρώπη μας ενδιαφέρει εκπρόσωποι όλων των χωρών, μεταξύ των οποίων και ε, η Σλοβακία, να μπορούν να μιλήσουν στην γλώσσα τους και ελπίζω ότι θα απαντήσετε στα σλοβακικά. Θαυμάσια λέει η πρόεδρος, η κυρία Σμόλκοβα. Ευχαριστώ πολύ. Εγώ θα μιλήσω σλοβακικά, στη μητρική μου γλώσσα. Κύριε Επίτροπε, άκουσα με μεγάλη προσοχή αυτά που είπατε Αναφέρατε στην παρέμβασή σας πάρα πολλά θέματα. Πράγματι, συνεχώς ακούμε πώς ανθιγίνα ζούνε, τρώνε και γενικά βιώνουν οι νέοι μας άνθρωποι. Ε, πόσο λίγο ασκούνται, ε, πόση λίγη άσκηση κάνουν και γενικά πόσο ανθιγίνα ζούνε με, δεν ενδιαφέρονται για τον αθλητισμό, για τα μαθήματα γυμναστικής, γενικά δηλαδή η άσκηση και οι ώρες ε, τις οποίες περνούν ασκούμενοι είναι, έχει μια φθήντουσα πορεία. Θα ήθελα λοιπόν να τονίσω ότι ε, έχει, πρέπει να κρούσουμε τον κόδωνα του κινδύνου, διότι ε, οι νέοι μας ε, δεν ασκούνται, δεν αθλούνται και πρέπει τουλάχιστον τρεις ώρες την εβδομάδα να διαθέτουν στον αθλητισμό. Ε, γι' αυτό λοιπόν θέλω να ρωτήσω τι σκοπεύει να κάνει η Κομισιόν, τι πρωτοβουλία σκοπεύει να αναλάβει για να μπορέσει να πραγματοποιήσει αυτό το αίτημα του αθλητισμού. Ο κύριος Τάκουλα, ευχαριστώ. θα είμαι σύντομο κύριε Επίτροπε, ε, αναφέρατε τη σημασία του εκπαιδευτικού προσωπικού. Υπάρχουν νέε πρωτοβουλίε για την κατάρτιση του εκπαιδευτικού προσωπικού στην Ευρώπη. Η κυρία Μπαντιά. Ευχαριστώ και ευχαριστώ κύριε Επίτροπε που ήρθατε σήμερα εδώ. Η σύμπτωση με τις δικές σας απόψεις και τις δικές μου είναι απόλυτη. Όντω, αυτά είναι τα θέματα που μα απασχολούν εμά εδώ στην Επιτροπή Πολιτισμού. Έχω όμω κάποιε συγκεκριμένε ερωτήσει. γιατί συμφωνούμε απόλυτα για το ότι πρέπει να βελτιωθεί η κατάρτιση. Όμω δεν φτάνει. Πρέπει την κατάρτιση αυτή να τη συντονίσουμε με την προσφορά εργασία. Γιατί βλέπετε ότι τα παιδιά που σήμερα είναι στο σχολείο ή φοιτητέ είναι αυτοί που μεθαύριο θα είναι στην αγορά εργασία. Έπειτα για την καινοτομία. Εκεί δεν πρέπει να προσανατολίσουμε την κατάρτιση των μαθητών και φοιτητών. Έχουμε και τη διαδικασία της Κοπεχάγης. Δεν πρέπει να λάβουμε υπόψη μας λοιπόν την καινοτομία, τη δημιουργικότητα, ώστε να έχει ο κόσμος ανοιχτό πνεύμα, ώστε να μπορεί να προσαρμόζεται στις αλλαγές της αγοράς εργασίας. Έπειτα είμαστε σε κρίση. Έχουμε νέους τομεί στην οικονομία, την πράσινη οικονομία. Μιλάμε για πράσινη απασχόληση. Φροντίζουμε να δώσουμε στους φοιτητές μας και τους μαθητές μας κατάλληλη κατάρτιση ώστε να μπορούν να είναι οι κατάλληλοι για αυτές τις νέες πράσινες θέσεις εργασίας. Αυτό με απασχολεί εμένα, το άμεσο μέλλον. Και θέλω να σας ρωτήσω κάτι και για την πρωτοβουλία που πάει φαντάζομαι προς αυτή την κατεύθυνση, το New Skills for New Jobs πώς θα προσαρμόσουμε την ε, εκμάθηση στις ανάγκες της νέας αγοράς εργασίας. Ωραία, λέει η Πρόεδρος, να μην ακούσουμε άλλη ερώτηση αυτή τη στιγμή για να δώσουμε την ευκαιρία να απαντήσει ο Επίτροπος. Θα ήθελα μόνο να πω ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση σε όλα αυτά τα ζητήματα μπορεί να δράσει μόνο επικουρικά. Κύριε Επίτροπε, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε. Και ευχαριστώ τα σχόλια της κυρίας, την κυρία Τρουιπέλ για τα σχόλια της. Όπως είπατε, θα πρέπει πραγματικά να φροντίσουμε για τη ε, νέα γενιά και να βρούμε ευρωπαϊκές λύσεις το, το, το, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο με την Κομισιόν πιστεύω θα προωθήσει όλα αυτά τα ζητήματα του χρόνου. Όσον αφορά την ε, διαβίου εκπαίδευση, είναι μια μεγάλη πρόκληση και συμφωνώ ότι χωρίς μια σωστή αναθεώρηση του προϋπολογισμού δεν θα μπορέσουμε να διαθέσουμε περισσότερες πιστώσεις σε αυτό τον τομέα ε, και να ε, αυξήσουμε τα κονδύλια, διότι εάν αναλύσουμε τα συν και τα πλην του προγράμματος από τη Γενική Διεύθυνση, διαπιστώνουμε δύο περιοριστικά στοιχεία. Πρώτον, τα χρήματα, τα κονδύλια, είναι προφανές περισσότερα χρήματα, περισσότερες ε, ενέργειες, περισσότερες δράσεις ε, περισσότερα προγράμματα, περισσότεροι συμμετέχοντες και περισσότερη συμμετοχή των νέων ανθρώπων και μάλιστα από φτωχότερα οικονομικο-κοινωνικά στρώματα. Θα είναι πραγματικά εντυπωσιακό πολλές φορές τι μπορούμε να επιτύχουμε με σχετικά μικρά κονδύλια. Μπορούμε να προβάλλουμε την τοπική, τον τοπικό πολιτισμό, την τοπική κουλτούρα, να την ε, ε, διαδώσουμε και πιο πέρα σε μεγαλύτερες περιφέρειες. Είναι λοιπόν πολύ σημαντικό να γίνει μία διαβούλευση συντονισμένη και να τονίσουμε ότι θέλουμε να επενδύσουμε σε, αυτές, σε αυτούς τους τομείς στο μέλλον. Θέλουμε να επενδύσουμε στη δημιουργικότητα, στην κατάρτιση και αυτά δεν μπορούν να γίνουν χωρίς τα, τις απαραίτητες πιστώσεις. Και κάτι ακόμα για το ε, Europeana είναι σαφές ότι έχουμε επιτύχει πολλά πράγματα με ένα σχετικό περιορισμένο, ε, σχετικά περιορισμένο προϋπολογισμό. Η Γεροπεάνα έχει μία βάση δεδομένων 4,7 εκατομμυρίων ε, πώς να θεμάτων, δεν είναι στοιχείων, δεν είναι μόνο εικόνες, φωτογραφίες, βιβλία, αλλά και άλλα στοιχεία τα οποία περιλαμβάνονται στην τράπεζα δεδομένων. Παραδείγματο χάρη αυτή η ψηφιακή βιβλιοθήκη του Google. Εάν λοιπόν τώρα πατήσεις ε, το πλήκτρο στο Google και Mozart, μία, ένα συνθέτη, έχεις χιλιάδες πληροφορίες ακόμα μπορείς να δεις στην οθόνη σου το πιστοποιητικό γέννησης του συνθέτη. Λοιπόν, πρέπει να βρούμε τρόπους πώς θα διατηρήσουμε και θα ε, ε, παγιώσουμε αυτό το μεγάλο επίτευγμα. Συμφωνώ μαζί σας 100%. Είναι σαφές ότι οι στόχοι, φιλοδοξίες ε, που έχουμε για την κινητοποίηση των τοπικών προγραμμάτων δεν μπορούν να καλυφθούν μόνο από ευρωπαϊκό προϋπολογισμό, αλλά πρέπει να συμβάλλουν και τοπικοί περιφερειακοί προϋπολογισμοί, επίσης ο ιδιωτικός τομέας μπορεί να συμμετάσχει οικονομικά στην Ευρώπη. Έχουμε μια μεγάλη παράδοση χρηματοδότηση προγραμμάτων από ιδρύματα, όπως παραδείγματο χάρη στις Ηνωμένε Πολιτείες. Εδώ πρέπει να πιέσουμε ε, περισσότερο, να διευρύνουμε τη συμμετοχή, την οικονομική στήριξη από αυτά τα ιδρύματα, τους οργανισμούς και τις ενώσεις. Όσον αφορά τον αθλητισμό, συμφωνώ μαζί σας. Ήμουν φανατικός ε, αθλητής στα νιάτα μου. Θυμάμαι πάρα πολύ καλά τι θαυμάσια αίσθηση είναι συμμετοχή σε μια αθλητική ομάδα, σε ένα σπορ. Είναι κάτι το οποίο ε, τα παιδιά σας θυμούνται για όλη τους τη ζωή. Δημιουργεί κοινωνικές σχέσεις, δημιουργεί το αίσθημα της, ε, της, ε, του, του, να ανήκει σε, μια ομάδα της φιλίας, της αλληλεγγύης. Γενικά δηλαδή ο αθλητισμός προσφέρει πάρα πολλά θετικά προσόντα στους νέους. Με τις νέες αρμοδιότητες πιστεύω ότι θα μπορέσουμε να εισάγουμε νέα στοιχεία στο αθλητικό πρόγραμμα. Και αυτά θα αναφερθούν στην ανακοίνωση την οποία θα προετοιμάσουμε την ερχόμενη εβδομάδα. Τώρα όσον αφορά την μητρική μου γλώσσα. Θα απαντήσω στη μητρική μου γλώσσα, στα σλοβακικά, με μεγάλη χαρά, μετά από αυτά που είπε ο κύριος Μιντόφσκι. Βεβαίως θα ήθελα να αναφερθώ και στην εργασία μας προς Ανατολάς. Η εταιρική μας σχέση προς Ανατολάς παρουσιάζει, προσφέρει ένα πολύ καλό παράδειγμα της διεύρυνσης και των θετικών επιπτώσεων της διεύρυνσης στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Έχουμε αυτή τη στιγμή συνάψει ε, νέες σχέσεις μέσα στο Σύμφωνο Συνεργασίας και Σταθερότητος με τις γειτονικές μας χώρες προς Ανατολάς, τις Ανατολικές και μέσα στη διαδικασία του LifeHub και ε, έχω, έχουμε αναπτύξει νέες ε, σχέσεις πιο σταθερές με την περιοχή των Βαλκανίων και αυτή τη στιγμή όλο το οικοδόμημα αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό από πλευράς δομικής, αρχιτεκτονικής πώς μπορούμε τώρα τα προβλήματα τα οποία έχουν χώρες μεταξύ τους ή και με εμάς να, τα, να τις βοηθήσουμε αυτές τις χώρες. Γι' αυτό ακριβώς ε, έγινε οργανώθηκε αυτή η πρωτοβουλία του Κίεβου και με τη διαδικασία αυτή θέλουμε να βελτιώσουμε τη συνεργασία της ε, και τις δομές αυτού του πλαίσιου, του εταιρικού πλαισίου και της γυτνίασης. Όσον αφορά τώρα την ανταλλαγή φοιτητών και εκεί θα προσπαθήσουμε να αναπτύξουμε αυτά τα προγράμματα μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των γειτονικών χωρών προς Ανατολάς και βεβαίως μέσω του προγράμματος Εράσμου, το οποίο προσφέρει μία παγιωμένη βάση στήριξης φοιτητών και δίνει τη δυνατότητα σε φοιτητές από όλο τον κόσμο να σπουδάσουν σε ευρωπαϊκά ιδρύματα, να αυξήσουν και να βελτιώσουν τις δεξιότητες τους, να αναπτύξουν το ταλέντο τους και πιστεύω ότι εργαζόμαστε προς αυτή την κατεύθυνση εξαιρετικά θετικά, με θαυμάσια αποτελέσματα και πιστεύω ότι η σημασία αυτών των προγραμμάτων θα αυξηθεί ακόμα περισσότερο στο μέλλον. Συμφωνώ και με την κυρία Σμόλκοβα, η οποία είπε ότι εάν κοιτάξουμε το α, παρελθόν, το, άμεσο παρελθόν, θα πρέπει να ανησυχήσουμε για την ε, έλλειψη ευκαιριών άσκησης και αθλητισμού. 42% των παιδιών, σύμφωνα με νέες μελέτες, κάθεται ώρες ατελείωτες μπροστά στην οθόνη ε, και δεν βγαίνει έξω ε, να παίξει όπως ε, παλιά, να σκηθεί, να τρέξει, να κάνει σπορ. Τα πράγματα έχουν αλλάξει από το παρελθόν. Δεν είναι μόνο τα παιδιά που κάθονται μέσα, αλλά και οι ενήλικες. Σε μία προφορική ερώτηση πρόσφατα πληροφορήθηκα ότι η κατανάλωση υδατανθράκων τη δεκαετία του 50 αυξήθηκε δραματικά και συνεχίζει να αυξάνεται λόγω της καθιστικής ζωής. Τι μπορούμε να κάνουμε προς αυτή την κατεύθυνση για να βελτιώσουμε αυτή την δυσμενή πραγματικότητα. Η Κομισιόν έχει συντάξει πολλά προγράμματα για, για τα σχολεία βάσει μιας ευρωπαϊκής στρατηγικής. Έχουμε το πρόγραμμα Νεότητα και Δράση, Youth and Action, η οποία στοχεύει στην ε, συμμετοχή των νέων πρέπει βεβαίως τα προγράμματα αυτά συνεχώς να προβάλλονται για να μην ξεχαστούν, έτσι ώστε να προσφέρουμε συνεχώς κίνητρα συμμετοχής των νέων σε αθλητικές ε, δραστηριότητες. Όσον αφορά τώρα την εκπαίδευση των ε, δασκάλων, πρέπει να πω ότι και σε αυτήν την περίπτωση πρέπει να ε, αποκτήσει την χαμένη του έγκλη το επάγγελμα και το λειτουργήμα ε, των ε, δασκάλων και των εκπαιδευτικών. Σε μερικές περιπτώσεις και σε ορισμένες χώρες έχουμε δυσκολία να στελεχώσουμε τα σχολεία. Έχουμε έλλειψη νέων που να θέλουν να γίνουν εκπαιδευτικοί. Ε, επίσης θα πρέπει ε, και έχουμε ήδη αναλάβει δραστηριότητες και πρωτοβουλίες έτσι ώστε να αυξηθεί η κινητικότητα των ε, δασκάλων. Πρέπει οι δάσκαλοι, οι εκπαιδευτικοί να ταξιδεύουν σε όλη την Ευρώπη, να βλέπουν τις βέλτιστες πρακτικές, να ανταλλάσσουν απόψεις με άλλους συναδέλφους, να μαθαίνουν τι γίνεται στις άλλες χώρες. Και πρέπει να συνεχίσουμε στην πορεία αυτή, γιατί πιστεύω ότι θα πρέπει να διδάξουμε τους δασκάλους πώς θα διδάσκουν σωστά τους νέους ανθρώπους, γιατί εκεί έγκυται και η επιτυχία του συστήματος στο μέλλον. Ευχαριστώ πολύ. Έχουμε άλλους έξι εγγεγραμμένους, ε, κύριο Σκούρια. Ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε. Πρώτα απ' όλα θα ήθελα πραγματικά να ευχαριστήσω τον ε, κύριο Επίτροπο, όχι μονάχα για όσα μας είπε σήμερα το πρωί, αλλά όπως και θα σας εξηγήσω καλύτερα σήμερα το απόγευμα, ε, για την μεγάλη του βοήθεια ε, στο θέμα του εθελοντισμού. Μας έδωσε όλα τα στοιχεία και τις δυνατότητες ώστε το Κοινοβούλιο να παίξει πρωταγωνιστικό ρόλο στο θέμα αυτό και θα ήθελα να τον ευχαριστήσω θερμά. Στην ερώτησή μου τώρα, ε, Πολλοί πιστεύουν ότι η εργασία στην Επιτροπή μας ε, είναι η καλύτερη και η ωραιότερη και εγώ πιστεύω όμως ότι δεν είναι μόνο αυτό, αλλά είναι και μια Επιτροπή της οποίας ε, το έργο είναι εξαιρετικά σημαντικό για το μέλλον της Ευρώπης. Ε, εγώ θα ήθελα λοιπόν να καταλάβω ποιες είναι οι στρατηγικές που η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και προκειμένου ο Επίτροπος προτίθενται να αναλάβουν έτσι ώστε ε, να ε, υπάρξουν περισσότερα κονδύλια ε, για να υλοποιηθούν οι ιδέες και επίσης ε, ποια είναι τα προγράμματα ε, τα οποία ε, προσβλέπουν την αύξηση της χορηγίας, στην ανάπτυξη του θεσμού της χορηγίας που είναι θεσμός απαραίτητος για την εξέλιξη του πολιτισμού. Η κυρία Μεναράπ. Κύριε Επίτροπε, κυρία Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι, σας ευχαριστώ πολύ για αυτή την ανταλλαγή απόψεων την οποία θεωρώ εξαιρετικά ενδιαφέρουσα. Θα ήθελα να θέσω το εξής ερώτημα πριν εκπαιδεύσουμε τα παιδιά μας έτσι ώστε να είναι έτοιμα για να εργαστούν, για να μπουν στην ε, αγορά εργασίας, δεν θα ήταν απαραίτητο να τους δώσουμε μία σημαντική βάση η οποία θα αφορά την καλλιτεχνική, γλωσσική και αθλητική εκπαίδευση και δεν θα έπρεπε ε, επίσης να αναπτύξουμε καλύτερα τα γνωστικά εργαλεία ε, έτσι ώστε να επιτρέψουμε στα παιδιά μας να είναι καλύτερα εφοδιασμένα όταν θα μπουν στην αγορά και στην πραγματική ζωή. Η πληροφόρηση είναι πάρα πολύ σημαντική οι πληροφορίες ε, που βρίσκουμε μέσα από το διαδίκτυο είναι σημαντικές, αλλά όπως είπατε και εσείς ε, υπάρχει τέτοια πληθώρα ε, πληροφοριών που πραγματικά μερικές φορές δεν ξέρουμε πώς να τις χρησιμοποιήσουμε. Άρα, πώς μπορούμε να διαχειριστούμε αυτόν τον μεγάλο όγκο πληροφοριών, πώς μπορούμε να τις ξεδιαλέξουμε, πώς μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τις πλέον κατάλληλες ε, και να τις χρησιμοποιήσουμε έτσι ώστε να αποκτήσουμε εφόδια ε, σαν πολίτες και σαν μελλοντικοί εργαζόμενοι. Ο προσανατολισμός, ο επαγγελματικός προσανατολισμός επίσης ε, είναι βεβαίως σημαντικός, αλλά εάν ξεκινήσουμε με έναν προσανατολισμό ο οποίος ε, θα γίνει σε πολύ πρώιμη φάση κινδυνεύομαι όταν τελειώσει το παιδί το σχολείο να έχει ξεπεραστεί πλέον ε, αυτός ο προσανατολισμός. Ζητώ συγγνώμη που δεν ε, μιλώ την δικιά μου μητρική γλώσσα αλλά είναι η γλώσσα των Βερβέρων η δικιά μου η οποία δυστυχώς εδώ δεν αναγνωρίζεται ως επίσημη γλώσσα. Ευχαριστώ πολύ κύριο Σανίσκη. Η κυρία Σανίσκη. Με μικρόφωνο παρακαλούμε. Για 45 χρόνια δουλεύω ε, ε, σαν τραγουδίστρια και καταλαβαίνετε ότι η δισκογραφική βιομηχανία της Ευρώπης ε, μου είναι ιδιαίτερος προσφυλής. Είναι μια ε, βιομηχανία όμως η οποία αυτή τη στιγμή διανύει ιδιαίτερα δύσκολη περίοδο, κυρίως λόγω της μουσικής πειρατείας γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά ότι μέσω αυτής της ε, πειρατικής πρακτικής ε, καταπατώνται όλα τα πνευματικά δικαιώματα. Και εδώ και πάρα πολλά χρόνια ε, δεν υπάρχει δυνατότητα να δοθεί μία δυνατότητα έτσι ώστε να λυθεί το θέμα αυτό. 52% των νέων τουλάχιστον ξέρουμε ότι χρησιμοποιούν την πειρατική πρακτική έτσι ώστε να κατεβάσουν μουσική και προγράμματα ε, online. Ε, όμως αυτό σημαίνει ότι τα προβλήματα δεν αφορούν μονάχα τους δημιουργούς αλλά και όλους ε, τους εργαζόμενους που ασχολούνται στον τομέα αυτό. Επομένως, ε, η, από τη στιγμή που δίδονται κονδύλια ε, και κρατικές επιδοτήσεις και κοινωτικές επιδοτήσεις έτσι ώστε να διατηρηθεί η ταυτότητα των ε, Ευρωπαίων δημιουργών, θα πρέπει να δοθούν κονδύλια και να, ώστε να προστατευτεί η μουσική και άλλη παραγωγή στην Ευρώπη. Ποια μέτρα λοιπόν προτίθεστε συγκεκριμένα να πάρετε κύριε Επίτροπε. Ευχαριστώ πολύ. Η κυρία Ναβετιλόβα. Θα ήθελα να συγχαρώ και εγώ, όπως οι προλαλήσαντες, τον Επίτροπο για την εξαιρετική σας παρέμβαση. Έχω μία ερώτηση που αφορά την ανταλλαγή φοιτητών από κράτη τα οποία είναι εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αναφέρεται το, την, ε, το πρόγραμμα Ευρωπαϊκής Συνεργασίας που δίνει αυτή τη δυνατότητα διαβλέπετε θετικές και ανωδικές τάσεις. Ε, πώς ε, εξελίσσεται η συνεργασία αυτή και οι ανταλλαγές με άλλες χώρες, με άλλες υπήρους όπως παραδείγματο χάρη από την Νότια Αμερική. Ε, είναι φοιτητέ που θέλουν να σπουδάσουν στα ευρωπαϊκά πανεπιστήμια τα οποία χαίρουν ιδιαίτερη εκτίμηση όπως αυτά και στι Ηνωμένε Πολιτείε. Ε, ε, πώς, τι σκοπεύει η Κομισιόν να κάνει για να προωθήσει τη διαβίου εκπαίδευση ώστε να μπορούν να ενταχθούν στα ειδικά προγράμματα. Elnök asszony, θα ήθελα και εγώ να ευχαριστήσω τον Επίτροπο. Πέρσι ήταν το έτος του διαπολιτισμικού διαλόγου και κατά τη διάρκεια αυτού του έτους ε, συνεργάστηκαν όλοι οι λαοί της Ευρώπης ε, και ε, οργανώθηκαν διάφορες εκδηλώσεις στο Βερολίνο γιατί είναι 20 χρόνια που έπεσε το τείχος. Όμως στη Γερμανία υπάρχουν ακόμα μεγάλες αντιθέσεις. Εχθές έγινε μια κρόαση με τις χώρες των Δυτικών Βαλκανίων για να προωθηθεί η συμφιλίωση ε, των λαών Ελπίζω να μπορέσει να επιτευχθεί η συμφιλίωση σε αυτό το μέρος των Βαλκανίων όπως έγινε και στη Γερμανία. Ε, τι μπορείτε να προσφέρετε προς αυτή την κατεύθυνση, παραδείγματος χάρη πρόθεση του διαλόγου των πολιτισμών, ε, της κουλτούρας, ε, των διαφόρων, διαφορετικών πολιτισμών μεταξύ ανατολικών και δυτικών περιφερειών, τι μπορείτε να κάνετε για την προώθηση της ευρωπαϊκής ταυτότητας. Και δεδομένου ότι μιλάμε για λαούς και γλώσσες, το νομοθετικό πλαίσιο για τη σλοβατική γλώσσα ακολουθεί λανθασμένη πορεία. πάρα πολλοί επιστήμονες και εμπειρογνώμονες της Σλοβακίας έχουν επικρίνει αυτό το νόμο. Ο Επίτροπος Μπαν, ε, ο οποίος είναι υπεύθυνος για την πολυγλωσία, δεν έχει σπείρει σωστό σπόρο. Καλά μίλησε για ε, την ε, πολυγλωσία, αλλά γιατί στη Ρουμανία, παραδείγματο χάρη, δεν υπάρχει πανεπιστήμιο που να διδάσκει στην ουγγρική γλώσσα ή λειτουργίες που γίνονται στα ουγγρικά. Και ε, είναι γεγονός ότι πολλά κράτη, πολλές κυβερνήσεις ακολουθούν ένα μονόδρομο όσον αφορά ε, την πολιτισμική και γλωσσική πολιτική. Εγώ πιστεύω για να προσεγγίσει η σλοβακική-ουγγρική συνεργασία θα πρέπει να γίνει μεγαλύτερη προσπάθεια να ανταποκριθούν στα αιτήματα των ε, εθνοτήτων που ζουν σε κάθε μία χώρα. Ε, οι, οι Σουηδοί, παραδείγματο χάρη, που ζουν στην Φιλανδία, χαίρον, ε, μπορούν να μιλήσουν ε, σουηδικά διότι αναγνωρίζεται η γλώσσα, έχουν μάλλον την, ε, το προνόμιο της μόρφωσης της παιδείας στα σουηδικά διότι αναγνωρίζεται ως επίσημη γλώσσα στη Φιλανδία τα σουηδικά. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε, κύριε Επιτροπή. Ήθελα και εγώ να θίξω το θέμα ε, των Αγγλικών και παρεμπιπτόν σας ευχαριστώ πολύ που μιλάτε Αγγλικά. είναι σημαντικό να μαθαίνει κανείς γλώσσες και υπάρχει μία αρχή που λέει ότι ε, καλό είναι τα παιδιά να μαθαίνουν, να διδάσκονται δύο επιπλέον γλώσσες πέραν της μητρικής τους και αυτό λειτουργεί σε ορισμένες ε, χώρες, σε ορισμένες άλλες δεν λειτουργεί τόσο καλά. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να μπορούμε να κατανοήσουμε ε, ο ένας τη γλώσσα του άλλου ε, και επομένως ε, να κατανοούμε καλύτερα ο ένας τον πολιτισμό του άλλου και είναι πολύ καλύτερο από το να υπάρχει μία μονάχα δεσπόζουσα γλώσσα. Το άλλο ζήτημα το οποίο θέλω να θίξω είναι ο αθλητισμός. Στην προηγούμενη θητεία του το Κοινοβούλιο συζήτησε σε βάθος το θέμα αυτό αλλά μερικές ε, φορές, ε, ε, ξέρετε όταν μιλάμε για αθλητισμό φέρνουμε στο μυαλό μας μονάχα το ποδόσφαιρο και μάλιστα την χρηματοδότηση μεγάλων ποδοσφαιρικών λεσχών. Νομίζω ότι θα πρέπει όταν μιλάμε για αθλητισμό να, μιλάμε, να μιλήσουμε για ένα πολύ πιο χαμηλό επίπεδο, δηλαδή για την δυνατότητα να αθλείται ο απλός κόσμος, για τη δυνατότητα να υπάρχουν αθλητικές εγκαταστάσεις οι οποίες θα είναι εύκολα προσβάσιμες ε, από όλους και όχι μονάχα για μεγάλα αθλητικά σωματεία κτλ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Χανιμπάλο. Ο κύριος Κέρκοπ. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Δύο πολύ σύντομα σημεία θα θίξω. Το πρώτο αναφέρεται σε αυτά που είπε η Μέρη πριν από δύο λεπτά. Ε, νομίζω ότι τη δεκαετία του 50 και του 60 όταν έγινε δημοφιλής η τηλεόραση ε, είχαμε, ξεκινήσαμε να έχουμε το πρόβλημα ότι πολλοί φίλεθλοι αντί να πηγαίνουν στι εθνικέ εγκαταστάσεις για να βλέπουν αγώνες να του παρακολουθούν από το σπίτι από την τηλεόραση. Ε, τώρα έχουμε ε, επίσης ε, την ίδια ε, αντιμετώπιση, δηλαδή ξαναρχίζουν οι νέοι να μένουν στο σπίτι τους, να μην αθλούνται, να μην πηγαίνουν στις, στις αθλητικές εκδηλώσεις, αλλά να τις παρακολουθούν από το σπίτι. Γενικότερα πάντως ο αθλητισμός είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό ο αθλητισμός ε, επίσης ε, είναι πολύ σημαντικό να είναι προσβάσιμος για ανθρώπους οι οποίοι δεν έχουν ε, κοινωνικό υπόβαθρο, εξαιρετικό ή οικονομικό υπόβαθρο. Οι άνθρωποι που μπορούν να αθλούνται είναι πάρα πολύ καλό να το κάνουν. Αλλά βλέπουμε ότι η ενθάρρυνση των ανθρώπων οι οποίοι δεν προέρχονται από κάποιο ε, ιδιαίτερα ψηλό κοινωνικό ή οικονομικό επίπεδο ε, είναι εξαιρετικά ε, σημαντικό ζήτημα. Και βλέπουμε ότι στον αθλητισμό σήμερα έχουμε πολλά τέτοια παραδείγματα. Επίσης να πω ότι ε, στην ε, ε, Ευρώπη ένα σημαντικό θέμα είναι τα δικαιώματα, τα πνευματικά δικαιώματα, όπως και τα δικαιώματα αναμετάδοσης. Θα πρέπει να προστατευτούν η πνευματική παραγωγή, η δημιουργία, τα τηλεοπτικά προγράμματα και αυτά θα πρέπει να τα προσέξουμε, γιατί είναι η προστασία των πνευματικών δικαιωμάτων είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Επίτροπο. Ο τελευταίος ομιλητής είναι ο κύριος Μπόρις. Ja również chciałbym życzyć powodzenia e, w Pana pracy, w ambitnych celach, które Pan stawia. Chciałem zwrócić uwagę... Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να κάνω δύο παρατηρήσεις. Πρώτο ε, θέμα η εκπαίδευση. Γνωρίζει ο κύριος Επίτροπος πολύ καλά ότι ειδικότερα στην κεντρική και ανατολική ε, Ευρώπη υπάρχουν ε, πολλά προβλήματα όσον αφορά αποκλεισμό ε, των υποψηφίων από ε, από πληροφορίες, έχουμε πρόβλημα όσον αφορά την πρόσβαση στο ίντερνετ, όσον αφορά την ευρυζωνικότητα. Ε, ελπίζομαι ότι τα επόμενα πέντε χρόνια μέσω χρηματοδοτήσεων θα ε, λήξει το πρόβλημα αυτό και επομένως θα είναι διαφορετική η κατάσταση όσον αφορά την πρόσβαση των Ευρωπαίων πολιτών, όλων των Ευρωπαίων πολιτών στην ευρυζωνικότητα. Ένα άλλο θέμα το οποίο θέλω να θίξω είναι η χρήση του διαδικτύου στην ε, διδασκαλία στα σχολεία, κυρίως ε, δε όταν ε, μιλάμε για μικρά σχολεία, για πόλεις ε, οι οποίες δεν, έχουν, ε, δεν δίνουν πολύ μεγάλες δυνατότητες και ευκαιρίες στους νέους. Αυτοί οι νέοι θα πρέπει να έχουν την δυνατότητα ε, να έχουν πρόσβαση στο διαδίκτυο, στην ευρυζωνικότητα, έτσι ώστε online να μπορούν να εκπαιδευτούν καλύτερα και να χρησιμοποιήσουν με τον βέλτιστο δυνατό τρόπο όλες τις πληροφορίες οι οποίες βρίσκονται στο διαδίκτυο. Να εκμεταλλευτούν δηλαδή τις νέες τεχνολογικές ε, δυνατότητες. Ε, αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό κατά την άποψή μου γιατί υπάρχουν πολύ μεγάλες ε, διαφορές στην Ευρωπαϊκή Ένωση όσον αφορά αυτό το, το ζήτημα και πιστεύω ότι αυτέ οι διαφορέ θα πρέπει να λήξουν. Ένα δεύτερο σημείο που ήθελα να θίξω είναι ο αθλητισμός που θα περιλαμβάνεται άλλωστε και στην συνθήκη της Λισαβόνας. Θα ήθελα ιδιαίτερα να σας ευχαριστήσω για αυτά που είπατε ε, για την ε, προσπάθειά μας ε, να καταρτήσουμε τους εκπαιδευτές που θα εκπαιδεύσουν τα παιδιά. Εγώ θα ήθελα να κάνω μια πρόταση όσον αφορά το θέμα αυτό. κυρίως δε όσον αφορά την ε, αθλητική εκπαίδευση σε όλα τα επίπεδα, μέχρι και το ε, επαγγελματικό. Ε, διαπιστώνουμε ένα ανησυχητικό φαινόμενο. Οι νέοι, οι οποίοι έχουν ταλέντο και οι οποίοι φτάνουν σε κάποιο υψηλότερο επίπεδο, πολύ συχνά αντιμετωπίζουν τεράστια προβλήματα πολλά προβλήματα στην επαγγελματική τους πλέον ε, ε, αποκατάσταση, δηλαδή στο να μπορέσουν να ασχοληθούν επαγγελματικά με τον ε, αθλητισμό. Και δεν αναφέρομαι μονάχα στο ποδόσφαιρο, αναφέρομαι και σε, σε όλα τα άλλα αθλήματα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση λοιπόν θα πρέπει να παρέμβει γιατί πολύ συχνά το μοναδικό κριτήριο όταν λαμβάνονται αποφάσεις ε, ε, το, το σημαντικό κριτήριο είναι τα χρήματα ε, και πολύ συχνά βλέπουμε εξοκοινοτικούς αθλητές οι οποίοι παίρνουν κατά κάποιο τρόπο τις θέσεις των Ευρωπαίων. Αυτό Σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. Ας προσπαθήσετε κύριε Επίτροπε να απαντήσετε. Ξέρω δεν μπορεί να απαντήσετε ενδελεχώς σε όλες τις ερωτήσεις αλλά έχετε την ευκαιρία τώρα να παρουσιάσετε τις απόψεις σας και τους επόμενους μήνες ελπίζουμε τη, να διατηρήσει τη θέση αυτή ένας άνθρωπος ο οποίος είναι τόσο εμπειρογνώμων και τόσο έμπειρος και, και τόσο ε, ικανός όπως ε, εσείς ε, και πιστεύω ότι αυτά όλα θα τα έχει υπόψη του ο Πρόεδρος της Κομισιόν, ο κ. Μπαρόσο. Λοιπόν, όσο μπορείτε πιο λεπτομερώς απαντήσετε. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Θα προσπαθήσω πράγματι να απαντήσω όλες αυτές τις ερωτήσεις όσο μπορώ πιο σύντομα. Σας ευχαριστώ πολύ λοιπόν για όσα μου είπατε, για την επικοδομητική σας προσέγγιση επίσης. Η δουλειά αυτή που γίνεται ε, για το έτος εθελοντισμού είναι όντως πολύ σημαντική. Συμφωνώ μαζί σας ότι τα προγράμματά μας πρέπει να διευρυνθούν περισσότερο. Πρέπει να δαπανάμε περισσότερα χρήματα και συγχρόνως να δαπανάμε καλύτερα. Άρα λοιπόν και στους δύο τομείς πρέπει να δουλέψουμε. Να δούμε τι περιθώρια υπάρχουν για να αυξηθούν τα κονδύλια που έχουμε στη θέση μας στο μέλλον και δεύτερον πώς μπορούμε τα κονδύλια αυτά να τα χρησιμοποιήσουμε καλύτερα. Και τα δύο. Η δικιά μου γενική διεύθυνση και εγώ ίδιος ξέρουμε πόσο σημαντικά είναι όλα αυτά τα προγράμματα στον τομέα της εκπαίδευσης, του πολιτισμού, του αθλητισμού. Έχουμε νέες ιδέες και τα στηρίζουμε προσπαθώντας να έχουμε περισσότερα κονδύλια στο μέλλον. Κάνουμε αξιολόγηση. Κοιτάμε αυτά τα προγράμματα, τι απέδωσαν στο εξωτερικό, ήταν αρκετά, ε, απέδωσαν όπως περιμέναμε καλύπτουν όλα τα κριτήρια, όλες τις προϋποθέσεις ώστε να θεωρείται επιτυχές ένα πρόγραμμα. Θα συνεχίσουμε να το κάνουμε αυτό και στο μέλλον. Με αυτή τη διτή προσέγγιση είμαι σίγουρος ότι θα γίνουμε πιο αποτελεσματικοί και θα έχουμε περισσότερα θετικά αποτελέσματα από τα προγράμματά μας αυτά. Νομίζω ότι στα γαλλικά τώρα με ρωτήσατε κάτι όσον αφορά την αναγκαιότητα κατάρτισης των ε, παιδιών πριν από το σχολείο. Είναι μια νέα ιδέα που την ε, ανακαλύψαμε τα τελευταία χρόνια. Καταλάβαμε δηλαδή τα τελευταία χρόνια ότι σήμερα το σύστημα εκπαίδευσης είναι πολύ απαιτητικό και γι' αυτό καλό είναι τα παιδιά να είναι ήδη προετοιμασμένα από πριν, όσο γίνεται πιο νωρί να αρχίσει η προετοιμασία αυτή. Βλέπετε, αν ξεκινάμε να μάθουμε ξένε γλώσσε νωρίτερα, συνήθω έχουμε καλύτερα αποτελέσματα. Συμφωνώ λοιπόν απόλυτα μαζί σας για το ότι σήμερα η ζήτηση είναι πολύ ευρεία, δηλαδή χρειάζονται διάφορες δεξιότητες, διάφορα προσόντα και είναι δύσκολο όλα αυτά να τα βάλουμε μέσα στο ίδιο κουρίκολο. Γι' αυτό και είναι πολύ σημαντικό να έχουμε ανταλλαγές βέλτιστων πρακτικών. Έχουμε τα κράτη, έχουμε σχολεία στα διάφορα κράτη, όπου διαπιστώσαμε εξαίρετα αποτελέσματα. Γι' αυτό λοιπόν είναι αναγκαίο να τη χρησιμοποιήσουμε την εμπειρία αυτή, να χρησιμοποιήσουμε δηλαδή πληροφορίες από το τι κάνουν οι άλλοι, έτσι ώστε να χρησιμοποιήσουμε τις καλύτερες δυνατόν προσεγγίσεις και αλλού. Προσπαθούμε να το κάνουμε αυτό μέσω του δικτύου μας Euridis, Ευρυδίκη, μέσω επίσης ε, μελετών που γίνονται και τα επόμενα χρόνια θέλω να πιστεύω ότι θα μπορέσουμε να αποφεληθούμε από τα πλεονεκτήματα των μελετών αυτών, από τα αποτελέσματα τα οποία μας δίνει το Ευρωπαϊκό Δίκτυο. Όπως επίσης και τα σχολεία τα οποία έχουν πετύχει πολύ στον τομέα της εκπαίδευσης για να προετοιμάσουν τα παιδιά σε διαφορετικού τύπου προσόντα. Έρχομαι τώρα στην κατάσταση όσον αφορά το διαδίκτυο. Έχετε απόλυτα δίκιο ότι τα μοντέλα συμπεριφοράς διαφέρουν από ό,τι ήταν πριν από μερικά χρόνια, σήμερα είναι εντελώ διαφορετικά. Γι' αυτό κάνουμε πολλές προσπάθειες, αυτό που ονομάζουμε αλφαβητισμό στο διαδίκτυο. Θέλουμε δηλαδή να φροντίσουμε, να μάθουμε στα παιδιά πώς μπορούν να δουλεύουν με το διαδίκτυο, τι μπορούν να κάνουν με τις πληροφορίες που υπάρχουν, πώς να τις ψάξουν. Είναι κάτι αρκετά καινούριο. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θέλει να επενδύσει πολλές προσπάθειες σε τέτοιου είδους προγράμματα για τη χρήση του διαδικτύου. Το κέντρο για ασφαλές διαδίκτυο που υπάρχει σε όλες τις χώρες μέλη, αυτό ακριβώς κάνει. Μπορεί κανείς να επικοινωνήσει με το κέντρο αυτό, να έχει ανταλλαγέ απόψεων με αυτό, ώστε να βελτιώσει την προετοιμασία των παιδιών στο διαδίκτυο. Έρχομαι τώρα στα, στο copyright και στα δικαιώματα των συγγραφέων και των καλλιτεχνών. Εδώ έχουμε ένα νέο τοπίο. Είπα ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή γνωρίζει πολύ καλά το πρόβλημα και πρέπει να προσπαθούμε να έχουμε μια ισορροπημένη λύση, μια ισορροπημένη προσέγγιση, ώστε να διασφαλίσουμε και τους τραγουδιστές, τους καλλιτέχνες, τους συγγραφείς, ώστε να παίρνουν την αμοιβή που τους πρέπει γιατί είναι ένας πολύ σημαντικός τομέας ευρωπαϊκού πολιτισμού και πολύ σημαντικός και για την ευρωπαϊκή οικονομία. Οπότε η επόμενη επιτροπή σίγουρα θα έχει μία διαβούλευση με όλους τους εμπλεκόμενους ώστε να πετύχει την ισορροπία αυτή. Όπως είπα και πριν, προστασία των εσόδων των δημιουργών, αλλά συγχρόνως διασφάλιση και της πρόσβασης του Ευρωπαίου πολίτη στον πολιτισμό. Είναι ξεκάθαρο ότι αυτό που θα προσπαθήσουμε να πετύχουμε ε, θα είναι κάτι το οποίο να είναι απλό, όχι περίπλοκο, όχι δύσκολο, που να μην εμποδίζει τους πολίτες να έχουν πρόσβαση στα πολιτιστικά αγαθά, από την άλλη μεριά θα φροντίσουμε να διασφαλιστεί και η σωστή αμοιβή των δημιουργών. Κατά τα άλλα. Και τώρα θα μιλήσω στη μητρική μου γλώσσα για τις ανταλλαγές των φοιτητών με μη ευρωπαϊκές χώρες. Πιστεύω ότι έχουμε επιτύχει πρόσφατα να σημειώσουμε μεγάλη πρόοδο σε, σε αυτό το ζήτημα μέσω του Εράσμους. Το πρόγραμμα αυτό έχει βελτιωθεί πολύ ε, οι υποτροφίες τώρα είναι συγκρίσιμες με τις υποτροφίες του Ιδρύματος Fulbright ε, και άλλα, άλλες υποτροφίες Αμερικανικών Ιδρυμάτων. Έχει αυξηθεί αριθμός των φοιτητών που συμμετέχει και υπάρχει και πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον για αυτό το πρόγραμμα. Ο προϋπολογισμός Άμα δείτε το προϋπολογισμό, ε, θα προσέξετε ότι μεγάλη προσοχή δίδεται σε αυτό τον τίτλο του προϋπολογισμού και παραμένει ένα πολύ σημαντικό ε, ε, πρόγραμμα προς χρηματοδότηση και στο μέλλον. Για τη διαβίου κατάρτιση πιστεύω ότι αυτός είναι ένας τομέας ο οποίος έχει προσλάβει ιδιαίτερη σημασία τον τελευταίο καιρό και πολύ περισσότερα κονδύλια έχουν εισρεύσει, αλλά πρέπει ακόμα, χρειαζόμαστε ακόμα περισσότερα. Οι στατιστικές μας λένε ότι σε 10 χρόνια η αργόρα εργασίας για άτομα με χαμηλές δεξιότητες, με λίγες δεξιότητες ή χαμηλής, ε, με χαμηλά προσόντα θα μειωθεί. Γι' αυτό και αυτό επειδή καταβάλουμε προσπάθειες αύξησης των προσόντων, βελτίωσης της κατάρτισης, έτσι ώστε τα άτομα να έχουν περισσότερες δεξιότητες. Υπάρχουν κατάλληλα προγράμματα τα οποία ήδη εκτελούνται ε, μέσα στα σχολεία ή εκτός των σχολείων. Δίνεται δηλαδή ευκαιρία, δεύτερη ευκαιρία κατάρτιση σε πολλούς ανθρώπους, ενήλικες κλπ. Και όσον αφορά τώρα τις διαφορές μεταξύ Ανατολής, Δύσης και και την κατάσταση μεταξύ παλαιότερων και νεωτέρων χωρών μελών. Κοιτάξτε τι έχουμε επιτύχει σε 20 χρόνια. Σε 20 χρόνια έχουμε επιτύχει εκπληκτικά πράγματα. Εχθές που βλέπαμε αυτά τα ντόμινο να πέφτουν στο Βερολίνο, κοιτάξτε στο, τι έχει γίνει στο τοπίο της Ευρώπης τα τελευταία 20 χρόνια. Τρομερά πράγματα. Το επίπεδο ζωής έχει βελτιωθεί, το επίπεδο της παιδείας, η μακροβιότητα, τόσα πολλά θετικά στοιχεία τόση πολύ πρόοδος που έχει επιτευχθεί και βεβαίως η ευρωπαϊκή ενσωμάτωση, η ολοκλήρωση της Ευρώπης. Βλέπετε λοιπόν πως οι δυτικέ χώρες έχουν, έχουν ωφεληθεί από τις ανατολικές χώρες, από τις νέες ε, δεξιότητες, δεξιότητες ε, το νέο πλούτο που εισέρχεται από τις καινούργιες χώρες. Like ε, και πώς έχουν αλλάξει τα πράγματα από αυτό που ήταν πριν από 20 χρόνια. Εάν δείτε τώρα τη μετάβαση από ένα απόλυτα πολιταρχικό σύστημα προς ε, την ε, πλήρη παγιωμένη δημοκρατία αυτών των χωρών, ε, πραγματικά είναι κάτι το εντυπωσιακό. Εγώ θυμάμαι όταν ήμουνα στο σχολείο έπεφτε το τείχος του ε, όταν ήμουν νεότερο έπεφτε, έβλεπα την πτώση του τείχους του Βερολίνου και τα παιδιά τώρα το μαθαίνουν σαν, σαν γεγονός της ιστορίας στο σχολείο. Και πραγματικά η πρόοδος της ε, ιστορίας ήταν ε, γεωμετρική. Μπορεί λοιπόν να είμαστε υπερήφανοι για την πολιτική συνοχή της Ευρωπαϊκής Ένωσης και, και με στοιχεία αλλά και με γεγονότα. Τα γεγονότα ήταν εντυπωσιακά. Όσον αφορά τώρα το γλωσσικό καθεστώς, η Κομισιόν είναι πολύ ικανοποιημένη από το θετικό γεγονός της ε, σύγκλησης ε, μεταξύ Σλοβακίας και Ουγγαρίας στο γλυκό ζήτημα. Είχαμε επανειλημμένες ε, συζητήσεις με τους αρμόδιους υπουργούς παιδείας αλλά και με τους υπουργούς εξωτερικών και υποσχέθηκαν οι δύο χώρες μέσα στα πλαίσια της ΔΑΣΕ και των μειονοτήτων να συνεργαστούν θετικά μαζί για να... Uh, uh, uh, Με στα πλαίσια της ΟΑΣΕ, συγγνώμη, να συνεργαστούν ε, έντονα για, την, ε, το γλωσσικό ζήτημα έτσι ώστε να μπορέσουν να καλυφθούν οι ανάγκες των μειονοτικών εθνοτήτων που ζουν στις δύο χώρες. Και πιστεύω ότι προς τα εκεί πρέπει να βαδίσουμε, να προωθούμε το διάλογο, καλές σχέσεις και να κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε για σχέσεις ε, καλής γυτνίασης, έτσι ώστε να υπάρχει ένα συνεχής ανοιχτός διάλογος προς κάλυψη των αναγκών και από τις δύο πλευρές. Αναφέρεται και τον Επίτροπο, ο οποίο είναι αρμόδιος για την πολυγλωσία, για το γλωσσικό καθεστώς μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Εάν αναλύσετε, αν δείτε ποια είναι τα εμπόδια ε, στους νέους τα οποία παρουσιάζονται όταν θέλουν να ε, εκμεταλλευτούν την ε, ενιαία αγορά, την, τα ανοιχτά σύνορα, συνήθως είναι το η γλώσσα. Η γλώσσα δημιουργεί προσκόμματα ελεύθερης κυκλοφορίας, εκπαίδευση και κατάρτιση σε άλλες χώρες, άρα δηλαδή σε άλλες γλώσσες. Γι' αυτό λοιπόν ο αρμόδιος επίτροπος δέχεται ότι η γλωσσική εκπαίδευση, οι, γλωσσική, γνώσεις πολλών γλωσσών είναι ένα μία απαραίτητη προϋπόθεση για την κινητικότητα των νέων και για να μπορέσουν να εκμεταλλευτούν τις ευκαιρίες που προσφέρουν οι ευρωπαϊκέ αγορέ. Επίση, οι ξένε γλώσσε, η εκμάθηση ξένων γλωσσών δημιουργεί γέφυρε προ άλλε χώρε, προ άλλου πολιτισμού και ανοίγει τις πόρτες στην κοινωνία της πληροφορίας, της ε, μιλώντας, το αναφερόμενο τώρα στα τηλεοπτικά δικαιώματα είναι όντως ένα λίαν περίπλοκο θέμα. Και γι' αυτό έχουμε ξεκινήσει έναν ευρύτερο διάλογο με τους ενδιαφερόμενους του τομέα και θα παρουσιάσουμε μια πρόταση πώς θα μπορέσουμε να διαχειριστούμε με τον καλύτερο τρόπο αυτόν τον τομέα των τηλεοπτικών δικαιωμάτων για να μπορέσουμε να υιοθετήσουμε τις καλύτερες προτάσεις, καλύτερες δηλαδή για όλους, για όλες τις πλευρές. Όσον αφορά το ε, διαδίκτυο και την εκπαίδευση μέσω του διαδικτύου, ήδη υπάρχουν προγράμματα σε αυτόν τον τομέα. Έχουμε πολύ θετική εμπειρία όσον αφορά τις ανταλλαγές μεταξύ σχολείων μέσω διαδικτύου, δηλαδή ε, ανταλλαγές ε, μάθησης ε, προγραμμάτων και γνώσεων στο σχολικό επίπεδο μέσω διαδικτύου και ο στόχος μας είναι να χρηματοδοτήσουμε την ευρυζωνική πρόσβαση σε όλη την Ευρώπη. Πραγματικά ελπίζω σε μερικά χρόνια να μην υπάρχει κανένα σημείο στην Ευρώπη που να μην έχει πρόσβαση στο ευρυζωνικό δίκτυο και τόσο αφορά τον αθλητισμό. Γνωρίζομαι πόσο σημαντικό είναι, πόσο σημαντικό είναι το ποδόσφαιρο για, για χώρες όπως είναι η Ισπανία, όπως είναι η Ιρλανδία, όπως είναι η Αγγλία, πόσο σημαντικό ρόλο παίζουν και ε, οι ποδοσφαιρικές ε, ομάδες. Αλλά πρέπει να σας πω ότι στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν ε, συζητάμε μονάχα για το ποδόσφαιρο ή για τις, με, με τα μεγάλα αθλητικά σωματεία, είτε μονάχα για τους πολύ μεγάλους φορείς του αθλητισμού. Εμάς μας ενδιαφέρει η πρόσβαση όλων των πολιτών ε, στον αθλητισμό ε, και ε, πραγματικά οι ιδέες σαν αυτές που αναφέρατε προηγουμένως είναι πάρα πολύ σημαντικές γιατί πραγματικά εμείς θα προσπαθήσουμε στη νέα ανακοίνωση της Επιτροπής να καλύψουμε τον επόμενο χρόνο, να καλύψουμε όλα τα θέματα σχετικά με τον αθλητισμό. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ κύριε Επιτροπή. Λέει η Πρόεδρος. Ευχαριστώ όλους όσους είχαν συμμετέσχον στη συζήτηση. Διαπιστώσαμε ότι τις, ε, τους επόμενους μήνες, τις επόμενες εβδομάδες έχουμε πάρα πολλά να κάνουμε σε πολύ διαφορετικούς τομείς. Από το copyright μέχρι τον αθλητισμό, από τη, τις επιχειρήσεις μέχρι τα πανεπιστήμια και πέραν αυτών στον εθελοντισμό, όλα αυτά τα οποία κάνουν τη ζωή μας ενδιαφέρουσα και ε, αξιόλογοι. Με όλα αυτά πρέπει να ασχοληθούμε. Έχουμε λοιπόν ένα πολύ σημαντικό έργο και ευχόμαστε η Κομισιό να μπορέσει να ανταποκριθεί σε αυτό το έργο της όπως έκανε και πάντοτε. Σας θυμίζω ε, και άλλους συναδέλφους που έχουν μιλήσει στο παρελθόν για τα, τις αρμοδιότητες κλειδιά τα οποία, πρέπει, τα, τα οποία έχει αναλάβει η Κομισιόν. Πράγματι, για αυτά τα κλειδιά μιλάμε τώρα. Είπαμε εξ ότι πρέπει να ξέρουμε ε, σαφώς τι πρέπει να γνωρίζει ένας νέος άνθρωπος, ε, τι γνώσεις πρέπει να έχει. Καταρχάς πρέπει να γνωρίζει πώς να αποκτήσει την ε, παιδεία που χρειάζεται. Να μάθει δηλαδή καταρχάς, να πληροφορηθεί πώς θα μάθει, πώς θα εκπαιδευτεί και μετά να τα βγάλει πέρα με τον Σέξπιρ ή τον Όμηρο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Επίτροπε. Ελπίζω να μπορέσετε να διατηρήσετε τη θέση σας. Έχετε ήδη ε, ενσωματωθεί θα έλεγα κατά εξαιρετικό τρόπο. Εάν, επιτύχει, εάν περάσετε τις εξετάσεις θα είναι μεγάλη χαρά για μας. Εάν όμως δεν τις περάσετε και ακολουθήσετε άλλη πορεία και εκεί είμαι σίγουρη ότι θα σημειώσετε μεγάλη επιτυχία λόγω των ε, ικανοτήτων σας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συνεργασία σας. Αγαπητοί συνάδελφοι, έχουμε τώρα μία πάρα πολύ ενδιαφέρουσα συνέχεια στην ημερήσια διάταξη. Και παρακαλώ όσοι συνάδελφοι έχουν κρυφτεί πίσω να έρθουν μπροστά στις θέσεις τους για να τους βλέπουμε. Ελάτε παρακαλώ στις πρώτες σειρές έτσι ώστε να μπορέσουν να καθίσουν στις πίσω στις θέσεις ε, οι διευθυντές, οι σκηνοθέτες των έργων που θα ε, συζητήσουν για τα βραβεία αυτά τα οποία θα δοθούν και τα οποία εκφράζουν την ευρωπαϊκή ψυχή, το ευρωπαϊκό πνεύμα. Λοιπόν, οι σκηνοθέτες και οι αρμόδιοι για τα, τα έργα θα κάτσουν σε μία πλευρά, αλλά θέλω τα μέλη μας να φαίνονται, να είναι ορατά. Θα διακόψουμε για δύο-τρία λεπτά που να κάτσουν όλοι. Okay. Ich spreche Deutsch. Wir sind ein multilinguales Parlament. So. Είμαστε πολύ γλωσσο σώμα, πολύ γλωσσο κοινοβούλιο. Καλωσορίζω λοιπόν, λέει η πρόεδρο, θερμά τους καλεσμένους μας. Η Αντιπρόεδρος κυρία Ντουράν είναι εδώ, χαίρομαι ιδιαίτερα μαζί με την Επιτροπή μας, Επιτροπή Πολιτισμού και Παιδείας, είναι ε, αρμόδια για την διεκπαιρέωση, τη σωστή διεκπαιρέωση της διαδικασίας του βραβείου Λουξ. Έχουμε αυτή τη στιγμή, φέτος δηλαδή, μία επιλογή θαυμάσια, τόσο καλή όσο δεν είχαμε ποτέ στο παρελθόν. Και γι' αυτό σας παρακαλώ μην ξεχνάτε ότι έχουμε και αίθουσα προβολή στον τρίτο, όροφο πίσω από το Vox Box όπου μπορείτε, υπάρχει ένα πρόγραμμα, ε, να δείτε τις ταινίες, τις υποψήφιες ταινίες. Ε, υπάρχουν ειδικέ ώρες προβολής των διαφόρων ταινιών, μεσημέρι, απόγευμα, βράδυ. Αλλά μπορείτε να το δείτε και μέσω του ειδικού καναλιού στο διαδίκτυο του Κοινοβουλίου. Αν δεν προλάβετε να τις δείτε εδώ. Αυτό αυτό το βραβείο Λουξ δίδεται, απονέμεται για, σε έργα, σε κινηματογραφικές ταινίες, οι οποίες έχουν ευρωπαϊκά θέματα. Και το βραβείο αυτό αποφασίζεται από, ένα ανεξάρτητο, από μια ανεξάρτητη επιτροπή βράβευσης και τα τρία, οι τρεις ταινίες που έχουν επιλεγεί προβάλλονται, μπορούν να, μπορείτε να τις δείτε, να τις παρακολουθήσετε και προβάλλονται δωρεάν και σας παρακαλώ πραγματικά να δείτε αυτά τα αξιόλογα έργα τα οποία αντανακλούν την ψυχή της Ευρώπης. Έχουμε εισαγάγει αυτή αυτό το βραβείο η ιδέα ήταν ε, του προηγούμενου αντιπροέδρου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ο οποίος πίστευε ότι κατά αυτόν τον τρόπο προβάλλεται καλύτερα το πνεύμα και η ψυχή της Ευρώπης. Και δεν πρέπει, πιστεύω, ε, τα έργα αυτά να μην ε, βλέπονται από τον κόσμο, να μην προβάλλονται και γι' αυτό είμαστε ιδιαίτερα ευτυχείς που έχουμε τη δυνατότητα να προβάλλουμε αυτές τις ταινίες και να τις δείτε διότι περιλαμβάνουν θέματα τα οποία μας απασχολούν στο σώμα, περιλαμβάνουν δηλαδή θέματα ευρωπαϊκής πολιτικής τα οποία μας έχουν απασχολήσει και θα μας απασχολήσουν. Στις 24 Νοεμβρίου στο Στρασβούργο θα δοθεί ε, το βραβείο στον νικητή και ε, το βραβείο αυτό δεν είναι χρηματικό, αλλά τα χρήματα αυτά θα χρησιμοποιηθούν για να υποτιτλιστούν υποτιτλιστεί η ταινία που θα βραβευτεί στις ευρωπαϊκές γλώσσες από την ε, ε, Ιρλανδία μέχρι τη Σλοβενία θα, μπορέσει, θα μπορέσουν οι θεατές να δουν τη ταινία αυτή υποτιτλισμένη στη γλώσσα τους. Το πρώτο βραφείο δόθηκε το 2007 στην ταινία ε, με γερμανικό τίτλο «Στην άλλη πλευρά». Και ο σκηνοθέτης... Σκηνοθέτης δεν είναι. Τι λέμε, παραγωγός ή σκηνοθέτης. Α, ωραία, ωραία σκηνοθέτης και παραγωγός. Δεν ξέρω ακριβώ την ορολογία, λέει η πρόεδρο. Και οι δύο είναι παρόντε και βεβαίω οι πρωταγωνιστές είναι εδώ μαζί μας και γι' αυτό χαιρόμαστε ιδιαίτερα. Καλωσορίζω την Χάνα Σιγκούλα, η οποία ε, έπαιξε έναν σημαντικό ρόλο σε αυτό το έργο και με τον ε, σκηνοθέτη βρίσκεται εδώ. Χαίρομαι επίσης που είναι εδώ ο κύριος Μέρκ, και ο Φάτι Ιακίμ, Ακίμ, ο οποίος έχει παρουσιάσει ένα καινούριο έργο φέτος. Ο Φατή Ακίν λοιπόν που κέρδισε το βραβείο αυτό το 2007. Χαίρομαι λοιπόν που οι τρεις ε, σημαντικοί ε, δημιουργοί, δηλαδή η πρωταγωνίστρια, ο σκηνοθέτης και ο παραγωγός ε, του πρώτου βραβείου που δόθηκε, της πρώτης βραβευμένης ταινίας, είναι εδώ σήμερα. Και έχουμε πραγματικά τώρα εμπειρία της μεγάλης αξίας αυτής, της, αυτού του βραβείου. και καλωσορίζω και τον αρμόδιο ο οποίος ε, φρόντισε να γίνει ο υποτιτλισμός της ταινίας αυτή σε 7 διαφορετικές γλώσσες. Είναι λοιπόν ένα θαυμάσιο υλικό αυτό στα χέρια μας, μια εξαιρετική ποιότητα ταινία με, σε 7 γλώσσες υποτιτλισμένη και τώρα έχουμε την καινούργια σοδιά ας πούμε των ε, δημιουργών Έχουμε μαζί μας τον Hans Christian Schmidt, ο οποίος είναι ο σκηνοθέτης της ταινίας ε, «Καταιγίδα», «Sturm» στα γερμανικά, «Καταιγίδα». Είναι ένα έργο το οποίο ε, ε, αναφέρεται στην εμπόλεμη εποχή της Βοσνίας. Και Έχουμε επίσης τον ε, σκηνοθέτη Καμέν Κάλεβ από τη Βουλγαρία που σε συμπαραγωγή με τη Σουηδία έχει ε, κάνει την ταινία Eastern Place, ανατολικά παιχνίδια. Ε, είναι λοιπόν του Καμέν Κάλεφ από τη Βουλγαρία η ταινία αυτή, μια πολύ δύσκολη ταινία που χειρίζεται ένα πολύ ευαίσθητο θέμα και Ορισμένοι συνάδελφοι από τη Βουλγαρία ε, ε, είπαν κάπως επιφυλακτικά πρέπει πάντοτε να δείχνουμε προβλήματα αρνητικά που αφορούν τη Βουλγαρία και είπαμε δεν είναι μόνο προβλήματα αυτά της Βουλγαρίας, είναι προβλήματα ολονών μας, ας είναι έστω και δυσάρεστα. Όλα πρέπει να αντιμετωπίσουμε. Ε, Επίση, υπάρχει μια άλλη ταινία αλλά δεν εκπροσωπείται από κανέναν εδώ σήμερα. Είναι το έργο Welcome στα αγγλικά, καλώς, ήρθατε, καλώς ορίσατε, ε, Γάλλου σκηνοθέτη του Φιλίπ ε, Λιωρέ. Ευχαριστώ λοιπόν ε, όλους τους δημιουργούς, παραγωγούς, συμπαραγωγούς που μας έκαναν την τιμή να έρθουν σήμερα εδώ. Σας καλωσορίζω και πάλι και σας σας παρακαλούσα να πάρετε το λόγο. Πρώτα ο κύριος Κάλεφ, μετά ο Φάτι Χακί, μετά η Χάνα Σιγκούλα και να κάνετε μια σύντομη παρέμβαση. Ε, να μας παρουσιάσετε δηλαδή σύντομα το, το, το, το έργο σας, την ταινία αυτή την οποία φτιάξατε πώς ε, έγινε αυτή η ταινία, ε, πώς μπορέσατε να λάβετε την απαραίτητη χρηματοδότηση και υποστήριξη, πώς οργανώσατε τη συγχρηματοδότηση, τι δυσκολίες αντιμετωπίσατε, πώς βρήκατε τους ηθοποιούς σας, γενικά δηλαδή την όλη διαδικασία δημιουργίας. Καταρχάς δίνω το λόγο στον κύριο Κάλεφ για πέντε λεπτά για να μας παρουσιάσει την ταινία του Eastern Plays. Κύριε Κάλεφ, έχετε το λόγο. Βουλγαρικά, γαλλικά, τι γλώσσα μιλήσετε. Είναι möglich? ναι. Οκ. Uh, uh, Ευχαριστώ. Μα αυτό ακριβώ είναι ένα από του λόγου για του οποίου χαίρομαι ιδιαίτερα μου που βρίσκομαι εδώ να παρουσιάσω αυτή τη βουλγαρική ταινία. Είναι μια ταινία που δείχνει λιγάκι την πραγματικότητα στις χώρες μας. Και είναι σημαντικό που προβάλλεται εδώ και σε διάφορες άλλες χώρες. Είναι πραγματικά πολύ θετικό, γιατί βλέπετε η ταινία αυτή στις μέρες μας είναι πάρα πολύ δύσκολο τέτοιου είδου ταινίε από μικρές χώρες όπως είναι η Βουλγαρία να έχουν την ευκαιρία να προβληθούν ευρέω. Αυτή λοιπόν είναι μια πολύ μεγάλη ευκαιρία για μας και είναι πολύ θετικό. Χρειαζόμαστε εικόνες για να δούμε αν υπάρχει ένα πρόβλημα ή απλώς και μόνο για να παρουσιάσουμε διαφορετικές απόψεις, διαφορετικές νοοτροπίες και να μπορούμε να μιλήσουμε για αυτά. Χαίρομαι λοιπόν που τόσος κόσμος μας παρακολουθεί και ότι τελικά θα υπάρχει η δυνατότητα να δείξουμε στο εξωτερικό το έργο μας. Πέρα δηλαδή από τη δικιά μας τοπική αγορά. Τώρα όσον αφορά την ταινία αυτή καθεαυτή, πρόκειται για κάποιους νέους που συναντάει κανείς παντού, ανά πάσα στιγμή, σε όλες τις χώρες, που έχουν τα ίδια προβλήματα, λίγο πολύ. Εδώ παίρνουμε το νεοναζισμό, αλλά μπορεί να είναι τα ναρκωτικά, μπορεί να είναι οτιδήποτε. Προβλήματα κοινά μεταξύ των νέων, μέσα στο οποία οι νέοι χάνονται, μπερδεύονται. και χάνουν την επαφή με τον ίδιο τους τον εαυτό, με την ταυτότητά τους. Σας ευχαριστούμε πολύ κυρικά. Αργότερα θα μπορέσουμε να συζητήσουμε και για άλλα θέματα. Σημείωσα τώρα, δεν θέλω να διακόψω τους ομιλητές, αλλά μετά, άμα θέλετε κάτι να ρωτήσετε, ευχαριστώ. Ο Hans Christian Schmidt έχει τώρα το λόγο. με κλειστό το μικρόφωνο, δεν τον ακούμε. Α, μικρόφωνο, ναι. Ευχαριστώ πολύ που μας προσκαλέσατε εδώ. Θα προσπαθήσω να πω στα αγγλικά και εγώ δύο λόγια. Η ταινία καταιγίδα και θα ξεκινήσω με την οικονομική πτυχή. Γιατί είπατε ότι θέλετε να ακούσετε και κάτι για τα οικονομικά. Λοιπόν, είναι μια γερμανο-ολλανδο-δανέζικη συμπαραγωγή. Με τον προπολογισμό χρειαστήκαμε Ευρωπαίους εταίρους, πήγε καλά. Η χρηματοδότηση ήταν φαντρίερη εταιρεία, η οποία ε, βοήθησε, ε, έψαξε στην Ολλανδία συμμετοχή και τελικά καταλήξαμε σε μια ιστορία που έχει να κάνει με το ποινικό δικαστήριο της Χάγης και την τέος Γιουγκοσλαβία. Γράφοντας το σενάριο καταλάβαμε ότι όπως συμβαίνει και εδώ στις Βρυξέλλες, ο καθένας μιλάει αγγλικά στο δικαστήριο. Οπότε καταλάβαμε ότι δεν είχε νόημα να συνεχίσουμε με το γερμανικό σενάριο, με γερμανούς ηθοποιούς, οπότε σκεφτήκαμε ότι μπορούσαμε να ψάξουμε να βρούμε καλύτερα διεθνείς ηθοποιούς. Γιατί στο ποινικό δικαστήριο υπάρχουν άνθρωποι από διαφορετικές χώρες που συνεργάζονται μεταξύ τους. Οπότε η αρχική γλώσσα δεν είναι μόνο τα αγγλικά, γιατί ορισμένοι είναι από την Κροατία, από την Βοσνία. Πάντως την εμπειρία τη βρήκα πάρα πολύ ενδιαφέρουσα για την ταινία αυτή καθεαυτή. Δεν ήξερα εγώ πολλά πράγματα για το ποινικό δικαστήριο στη Χάγη, ούτε ήξερα πολλά πράγματα για τον πόλεμο στα Βαλκάνια. Εγώ ήμουνα τη δεκαετία του 90 στη Δανία, ε, στη Φιλανδία. Α, συγγνώμη, σε ένα σχολείο στο Μόναχο που μάθαινα για ταινίες, να φτιάχνω ταινίες. Και τελικά έγραψα κάτι για έναν δικαστή στη Χάγη, γιατί ακριβώς είχα συναντηθεί με μία δικαστήνα και τελικά διαπίστωσα ότι ε, υπήρχαν και πράγματα για βιασμούς που είχαν γίνει. Και εδώ πρόκειται για μια γυναίκα η οποία είχε βιαστεί και που ήταν μια υπόθεση λοιπόν που είχε αναλάβει δικαστήνα αυτή που είχα γνωρίσει ε, για έναν βιασμό και προσπαθούσε να πείσει την ε, κοπέλα το θύμα να καταγγείλει τον βιασμό αυτό. Τώρα ασχολείται με την, τον Κάραζιτς, με την δίκη του Κάραζιτς η δικαστή αυτή. Ακούσατε ότι υπάρχει αναβολή μέχρι το Μάρτιο ίσως. Οπότε θα ετοιμάζεται στο μεταξύ η κυρία αυτή, η δικαστήνα. Πάντως δεν πρόκειται τόσο πολύ για ένα θέμα, πρόκειται περισσότερο για έναν άνθρωπο, για την ακαιρεότητα. Εδώ στην ταινία έχουμε δύο γυναίκες οι οποίες συναντιόνται κάποια στιγμή τη ζωής τους και πρέπει να αποφασίσουν αν μπορούν να συνεχίσουν σαν να μην έχει συμβεί τίποτα στη ζωή τους μετά από τα γεγονότα αυτά του πολέμου ή αντίθετα πρέπει κάτι να αλλάξουν. Και αυτό είναι το κέντρο της δουλειά μου. Είναι ο κόσμος, οι άνθρωποι, οι χαρακτήρες, οι προσωπικότητες πολύ περισσότερο από ότι δικαστήριο, πόλεμος. Δεν είναι αυτά τα αντικείμενα της ταινία μου, όχι. Είναι ή χαρακτήρες, για να Μαρία Μαρίνκα, ε, για παράδειγμα. Αυτά. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε. Φάτι Ακίμ, παρακαλώ, για πείτε μας κι εσείς για την ταινία και για το βραβείο Λουξ. Τι πιστεύετε. Μπορείτε να μας πείτε αν κατά πόσο χάρη στο βραβείο που πήρατε πέρυσι η ταινία σας ε, προχώρησε καλύτερα. Τους ελπίζω να έχετε να μας πείτε καλά πράγματα γι' αυτό. Ευχαριστούμε πολύ. Όλα τα ε, βραβεία τα οποία ε, παίρνει κανείς είναι πάρα πολύ σημαντικά. Καταλαβαίνετε ότι μια ταινία κινηματογραφική αφορά την επικοινωνία και επομένως αν ε, καταφέρουμε να περάσουμε το μήνυμα και να επικοινωνήσουμε και να ε, ε, μεταφέρομαι την, το, το μέλημα το οποίο μας έκανε να, κάνουμε την ταινία αυτή, τότε τόσο το καλύτερο και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Όσον αφορά το βραβείο, βεβαίως χαίρομαι, χαίρομαι πάρα πολύ. Αλλά παρόλα αυτά θα ήθελα να σας δώσω και μια συμβουλή για το μέλλον, αν μου επιτρέπετε καλό θα ήταν να δουλέψουμε περισσότερο με τις εικόνες. Η γλώσσα βεβαίως είναι κάτι εξαιρετικό, είναι ένα εξαιρετικό μέσο επικοινωνίας, αλλά εγώ ε, περνάω τώρα μία φάση ε, που θα ήθελα πιο πολύ να ασχοληθώ με, την, με τις εικόνες και με την επικοινωνία μέσω των εικόνων. Αυτά όσον αφορά ε, τη Ε, όσον αφορά ε, την, ταινία και το βραβείο. Τώρα, ε, σχετικά με την νέα ταινία, ξέρετε ότι είναι μια τριλογία για την αγάπη, για τον θάνατο και για το διάβολο. Αναρωτιέμαι πώς συνεχίζει τη ζωή του κάποιος ο οποίος έχασε ένα αγαπημένο του άτομο. Ε, η Χάνα Σιγκούλα έχει χάσει το γιο τη και επομένω πρέπει να δούμε πώς μπορεί να αντιμετωπίσει ένα τέτοιο σκληρό χτύπημα τη μοίρα. Μπορεί ε, ένα άνθρωπο ο οποίος έχει περάσει από αυτή τη διαδικασία, από το θάνατο, μπορεί να ξαναβρει το γέλιο, μπορεί να ξαναβρει τη χαρά της ζωής. Απ' την άλλη πλευρά μπορεί να περάσει δηλαδή αυτό το σύνορο και βεβαίως μετά αναφέρομαι και σε άλλα σύνορα, στα γεωγραφικά σύνορα ας πούμε. Ε, το σύνορο ανάμεσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και την Τουρκία. Η ταινία αναφέρεται σε μια καταδιοκόμενη ε, ε, πολιτική εξτρεμίστρια η οποία καταφεύγει στην Γερμανία ζητώντας άσυλο. Κοιτάξτε, η Τουρκία βεβαίω θέλει να γίνει ε, μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωση. Φυσικά έχει κάνει ένα αρκετά μεγάλο κομμάτι του δρόμου. Ε, και ε, επομένως έχει κάνει διάφορες προσπάθειες και επομένως η γερμανική πλευρά λέει «Μα κοιτάξτε, εμείς έχουμε δώσει ένα σωρό λεφτά ε, προσπαθώντας να βοηθήσουμε την Τουρκία να εκδημοκρατιστεί, να πάει προς το σωστό δρόμο, επομένως δεν μπορούμε να δώσουμε και άλλα χρήματα να ζητήσουμε από τους Γερμανούς φορολογούμενους έτσι ώστε ε, να, δώσουμε το, δώσουμε άσυλο σε αυτή την κυρία, την, επιστρέφουμε στο σπίτι της, τη γυρνάμε στο σπίτι της. Βεβαίως, μιλώντας για σύνορα μπορούμε να μιλήσουμε για άλλα σύνορα, μπορούμε να μιλήσουμε για τα σύνορα Μεξικού ε, Ηνωμένων Πολιτειών. Μπορούμε να μιλήσουμε για τα σύνορα ανάμεσα στον χριστιανισμό ε, και τον συντηρητισμό. Dahinter, auf der anderen Seite der Ideologien, da muss doch die Philosophie ε, είναι πολύ σημαντικό λοιπόν να βρούμε το φιλοσοφικό υπόβαθρο που ενώνει τους ανθρώπους πέρα από οποιασδήποτε διαφορές τους. Αυτό το φιλοσοφικό υπόβαθρο που αφορά στο θάνατο. Επιστρέφοντας λοιπόν στα πρώτα μου λόγια, λέω ότι η ταινία αφορά την επικοινωνία. Χάνα Σιγκούλα, θέλετε να πάρετε το λόγο. Θέλετε να μας ε, πείτε ποιες είναι οι εντυπώσεις, να μοιραστείτε μαζί μας κάποιες ε, ιδέες. Πώς είδατε τη συνεργασία σας. Ε? Ναι. Έχω κάνει πολλές ταινίες καλές, καλύτερες, λιγότερο καλές, πάρα πολύ καλές. Και μετά έκανε και αυτήν την ε, ταινία. Και πρέπει να σας πω ότι παρουσιάζει ένα ιδιαίτερο χάρισμα η ταινία αυτή. Ακόμα σήμερα με σταματάνε καμιά φορά στο δρόμο και μου λένε «Α, θυμάμαι την ταινία Α ή Β». Και δεν αναφέρομαι μονάχα στη Γερμανία, μερικές φορές στο Παρίσι, στο δρόμο με σταματάνε, με φιλούν. και σχεδόν βλέπω μια έκφραση ευγνωμοσύνης γιατί υπάρχει ε, μια ταινία οποιοδήποτε είδους μια ταινία η οποία σε επίπεδο ανθρώπινο ενδιαφέρεται ε, για τους ανθρώπους και αγγίζει τελικά τους ανθρώπους, γιατί αυτό είναι ο άνθρωπος, ο, είναι ε, ο άνθρωπος ο οποίος βρίσκεται αντιμέτωπος με τη ζωή και το θάνατο κάθε μέρα, που πρέπει να αντιμετωπίσει την απώλεια ενός αγαπημένου ανθρώπου. Όλοι όσοι βρισκόμαστε σήμερα εδώ είμαστε καλά, αλλά υπάρχουν προφανώς, αλλά υπάρχουν τόσοι άλλοι άνθρωποι οι οποίοι δεν είναι καθόλου καλά. Όταν είμαι στο Παρίσι βλέπω πόσοι άνθρωποι ε, ε, κοιμούνται στο δρόμο. Βλέπουμε ότι ο αριθμός τους διπλασιάζεται κάθε τόσο. Είναι οι άστεγοι, τον οποίων ο αριθμός διπλασιάζεται κάθε χρόνο. Πότε θα μπορέσουμε να σταματήσουμε ε, αυτή την κατάσταση. Πότε θα μπορέσουμε να περάσουμε το σύνορο αυτό. Και δεν πρέπει να δεχτούμε ότι υπάρχουν δύο, τρεις, τέσσερις κατηγορίες ε, ανθρώπων. Πρέπει να συνεχίσουμε να αγωνιζόμαστε και νομίζω ότι αυτή είναι και η κεντρική ιδέα όλων των επιλεγμένων ε, ταινιών. Δεν είναι δυνατόν να δεχόμαστε να μας λένε οτιδήποτε. Δεν είναι δυνατόν ε, να δεχτούμε ορισμένοι να ζουν όλο και καλύτερα, ενώ κάποιοι άλλοι ζουν όλο και χειρότερα. Και η ταινία του Φατή είναι μια πολύ προχωρημένη κίνηση. Δεν διαπίστωσε απλώς ότι κάτι δεν πάει καλά. Προχωράει ακόμα παραπέρα. Θέλησε να ε, δείξει μια, την ιστορία μιας γυναίκας και θα σας μιλήσω εδώ για το ρόλο μου λοιπόν μιας ε, γυναίκας ε, που στην αρχή δεν είναι ούτε πολύ καλά, ούτε ε, πολύ άσχημα, δεν είναι ούτε καλύτερο ούτε χειρότερο δηλαδή από το μέσο όρο των ανθρώπων, αλλά κάποια στιγμή αντιμετωπίζει μια καταστροφή και πρέπει να ξεπεράσει την προσωπική της ε, καταστροφή. Κάποια στιγμή στη ζωή μα όλοι είμαστε αντιμέτωποι με μια καταστροφή, οποιαδήποτε μορφή και αν έχει αυτή. Η γυναίκα αυτή όμως δεν γεμίζει με πικρία και καταφέρνει να κατανοήσει την άλλη πλευρά, την αντίπαλη πλευρά και προσπαθεί να προσφέρει κάτι αντί να ε, ε, γεμίσει πικρία, παράπονο και θλίψη. Οι συνθήκες που παρουσιάζονται στην ταινία είναι πολύ συγκεκριμένες. Αναφέρονται στη συγκεκριμένη περίοδο την ιστορική αυτής της περιοχής. Όμως μπορεί να μεταφερθούν και να ερμηνευθούν ότι συμβαίνουν και σε άλλες περιοχές του κόσμου, σε άλλες συνθήκες. Η ταινία αυτή, πόσες γλώσσες υπάρχουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση, 23-27 πάνω, θα υποτιτλιστεί ε, στις γλώσσες αυτές, όλες τις ευρωπαϊκές γλώσσες και αυτό είναι πολύ σημαντικό, διότι έτσι μπορούμε να καταλάβουμε καλύτερα ότι ζούμε σε διαφορετικούς κόσμους, αλλά όλοι είμαστε άνθρωποι. Το ανθρώπινο στοιχείο δηλαδή θα ε, υπερισχύσει ως νόημα αυτής της ταινίας. Η κυρία Πάκα ε, Ευχαριστώ την Χάνα Σιγκούλα και τώρα δίνω το λόγο στον εκπρόσωπο του Ινστιτούτου Γκέτε. Για να μας πει πώς θα βοηθήσει ακόμα περισσότερο στην προβολή της ταινία. Αφήστε το μικρόφωνο σας παρακαλώ για να μπορέσουμε και εμείς να προστατεύσουμε, να ακούσουμε καλύτερα. Ωραία, ωραία. Θα μιλήσω αγγλικά. Πρώτα απ' όλα πρέπει να παραδεχτούμε ότι για όλους εμάς ο κινηματογράφος ε, είναι ε, ένα πάρα πολύ σημαντικό μέσο επικοινωνίας ε, και λόγου και εικόνων. Μεταφέρεται και ο λόγος, ταξιδεύουν και οι εικόνες. Βλέπουμε ξένες ταινίες και μπορούμε να μελετήσουμε τα κοινωνικά φαινόμενα που υπάρχουν σε άλλες χώρες. Πρέπει όμως δυστυχώς να πούμε και να παραδεχτούμε ότι σε ορισμένες χώρες η εθνική κινηματογραφική ε, βιομηχανία είναι πιο σημαντική από ότι ε, κάποιες ε, άλλες παραγωγές. Στην Γαλλία, ας πούμε, βλέπουμε ότι ε, τα πράγματα είναι αρκετά καλά και υπάρχει ένα 30% εθνικής κινηματογραφικής παραγωγής, ε, αλλά σε άλλες χώρες ε, είναι δύσκολο να αντιμετωπίσει κανείς τον αμερικανικό κινηματογράφο. Είναι πάρα πολύ δύσκολο να δει κανείς βουλγαρικές ταινίες σε γερμανικούς κινηματογράφους και ελπίζουμε ότι στο μέλλον θα υπάρξουν περισσότερες, ανταλλα... θα περισσότερες ανταλλαγές ανάμεσα στις κινηματογραφικές βιομηχανίες των ε, χωρών. Ε, σε γενικές ε, γραμμές βλέπουμε μονάχα ταινίε υποτιτλισμένε στις μεγάλες χώρες. Δηλαδή δύσκολα βρέπει κανεί ταινία υποτιτλισμένη στα σλοβακικά και αυτή είναι μια πολύ μεγάλη ευκαιρία που μας δίνεται μέσω ε, του θεσμού των ε, βραβείων ε, Λουξ. Αυτός ο υποτιτλισμός λοιπόν σε 23 γλώσσες που έγινε μέσω του βραβείου Λουξ ήταν πάρα πολύ σημαντική ένα πάρα πολύ σημαντικό θέμα, μια πολύ σημαντική κίνηση. Επίσης είδαμε υποτιτλισμό στα κινέζικα, στα ινδονησιακά ε, κτλ. Ε, και με τον τρόπο αυτό ε, οι ευρωπαϊκές αξίες γίνονται γνωστές όχι μονάχα εντός των συνόρων της Ευρωπαϊκής Επικρατείας αλλά και εκτός και σε μερικές περιπτώσεις σε πολύ μακρινές ε, χώρες. Ε, αναφερόμαστε σε αξίες πολύ σημαντικές όπως είναι ε, η ανεκτικότητα, όπως είναι η δυνατότητα συμβίωσης. Μεταλαμπαδεύομαι λοιπόν κάποιες ιδέες οι οποίες ίσως είναι λιγότερο γνωστές σε ένα σημείο του κόσμου. Ευχαριστώ. Χαίρομαι λέει πρόεδρος, ότι το βραβείο Λουκ δίνει τη δυνατότητα να χρησιμοποιηθούν τα χρήματα αυτά κατά πολύ ε, χρήσιμο τρόπο, επικοδομητικό τρόπο και από άλλους. Εάν λοιπόν κατευθυνθούν προς την Ινδονησία, προς άλλες ε, περιοχές ε, του κόσμου, θα συμβάλλουν ακόμα περισσότερο στην διαπολιτισμική κατανόηση, διότι προσπαθούμε και εμείς να διευρύνουμε την ευρωπαϊκή διάσταση προσθέτοντας το, την παγκόσμια Europa ε, Mundus, την, προσθέτοντας το στοιχείο της παγκοσμιότητας και την παγκόσμια διάσταση στην ευρωπαϊκή. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την εισαγωγή σας, για την ε, ε, παρουσίασή σας και θα παρακαλούσα τους συναδέλφους τώρα να θέσουν ερωτήσεις σε μια μοναδική ευκαιρία που έχουμε σήμερα. Η κυρία Μπαντία, ακούσε πρώτα. Ευχαριστώ πάρα πολύ που ήρθατε σήμερα εδώ όλοι όσοι έχετε εμπλακεί σε αυτή την ωραία περιπέτεια. Μια στιγμή, μια στιγμή να βάλουν τα ακουστικά τους οι προσκεκλημένοι μας για να σας καταλαβαίνουμε, λέει ο Πρόεδρος. Εντάξει τώρα. Να, και τα ισπανικά, γιατί να μην βάλουμε και τα ισπανικά σε αυτήν την Βαβυλωνία, όπως την είπατε. Λοιπόν, έλεγα, ευχαριστώ που ήρθατε. Είναι το πρώτο βήμα ή ένα από τα πρώτα βήματα για να πάμε προς την ε, κατεύθυνση του ευρωπαϊκού κινηματογράφου. Γιατί όλοι ξέρουμε την αμερικανικός ε, κινηματογράφος, έτσι, τις ταινίες τη αμερικάνικες τις ξέρουμε όλοι πάρα πολύ καλά. Τι είναι όμως ο ευρωπαϊκός κινηματογράφος, είναι ο γαλλικός, ο αγγλικός, ο γερμανικός, ο δανέζικος. Ε, λοιπόν, αυτή η περιπέτεια που ξεκίνησε το 2007 με τα βραβεία Lux είναι το πρώτο βήμα ώστε να εξηγήσουμε τι είναι ο Ευρωπαϊκό κινηματογράφο. Γιατί οι ταινίε αυτέ για τι οποίε μιλάμε και που ακόμα δεν τι έχω δει φέτο, θα τι δω, αλλά έχουμε την εμπειρία να από αυτή την ταινία έχουμε εδώ τον σκηνοθέτη, τον παραγωγό, εξαιρετική ταινία και την ηθοποιώ. δείχνει ακριβώ τι είναι ο ευρωπαϊκό κινηματογράφο. Όχι ο κινηματογράφο μια χώρα, αλλά ευρωπαϊκό κινηματογράφο. Γιατί μιλά για ευρωπαϊκά προβλήματα, για ευρωπαϊκέ αξίε, για ευρωπαϊκέ νοοτροπίε και έτσι πιστεύω ότι έχουμε να προσθέσουμε κάτι στον ευρωπαϊκό πολιτισμό. Εμείς οι Ευρωπαίοι έχουμε κάτι ιδιαίτερο. Θέλουμε να βρίσκουμε την ταυτότητά μας βασιζόμενη σε αυτό που μας χωρίζει, όχι σε αυτό που μας ενώνει. Έχουμε διαφορετικούς πολιτισμούς, νοοτροπίες, γλώσσες, αλλά γιατί να μην κοιτάξουμε καλύτερα αυτό που μας ενώνει, αντί να κοιτάμε αυτό που μας χωρίζει. Γι' αυτό λοιπόν πιστεύω ότι η εμπειρία αυτή είναι πάρα πολύ καλή και ειλικρινά σας ευχαριστώ για τη δουλειά σας. Σας παρακαλούμε όμως και εσείς να βοηθήσετε εμάς. Πείτε μας, δείξτε μας, τι να κάνουμε, πού πρέπει να επενδύσουμε τα χρήματά μας, τι προσπάθειες πρέπει να κάνουμε, γιατί αυτός είναι ο καλύτερος τρόπος για να φροντίσουμε η Ευρώπη να προχωρήσει, να φτάσει μακριά και καλά. Ευχαριστώ. Η κυρία Ευχαριστώ, Ντόρις θα αρχίσω με μια προσωπική παρατήρηση γιατί η ταινία αυτή με τίτλο «Από την άλλη πλευρά» μου άρεσε τόσο πολύ διότι διαδραματίζεται στη Γερμανία και μάλιστα στη γειτονιά μου 200 μέτρα από τη γειτονιά μου. Και καταλαβαίνετε ότι αυτό είναι πολύ στην καρδιά μου μέσα όταν βλέπεις μια ταινία που αφορά τη γειτονιά σου. Επίσης μου άρεσε πάρα πολύ αυτή η ταινία διότι όπως είπατε ήδη η νέα πρωταγωνίστρια έχει μία ακραία προσέγγιση, πολλές φορές ε, μία έντονη αντιευρωπαϊκή ε, προσέγγιση κατά της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά τονίζεται επίσης την ε, στενή σχέση της Ευρώπης με άλλες χώρες όπως παραδείγματος χάρη την Κωνσταντινούπολη, και άλλες γειτονικές ε, πόλεις και, περιοχές, και κράτη και αυτό δείχνει ότι η πραγματικότητα ε, πολλές φορές είναι διαφορετική από την ιδεολογική βάση την οποία ασπαζόμεθα. Άλλο η ιδεολογία, άλλο η πραγματικότητα. Και ε, τις επόμενες μέρες θα δω βεβαίως ε, και τις ε, άλλες δύο ταινίες, αλλά σε πολλοί Ευρωπαίοι πολίτες έχουν παραστεί μάρτυρες αυτής της ακραίας αντιπαράθεσης και του εμφύλιου πολέμου που έγινε στην Βοσνία και στην περιοχή, η ευρύτερη περιοχή αυτή την Ευρωπαϊκή, ένας πόλεμος εξόντωσης δηλαδή. Και αυτά τα οποία συνέβησαν είναι ένα ε, βασίτατα ευρωπαϊκό πρόβλημα το οποίο ούτε έχει αναλυθεί επαρκώς, ούτε έχει βεβαίως ακόμα λυθεί απολύτως. Αποτελεί λοιπόν το θέμα της ταινία αυτής μια πολύ σημαντική συμβολή στο πρόβλημα στην ευρωπαϊκή διάσταση και στα προβλήματα τα οποία έχουν ε, επηρεάσει την Ευρώπη τις τελευταίες δύο δεκαετίες. Και η τελευταία παρατήρηση. Ο υποτιτλισμός στις ευρωπαϊκές γλώσσες είναι μία νέα πραγματικότητα η οποία μόνο κέρδος θα αποφέρει. Είναι δηλαδή μια κατάσταση όπου θα κερδίσουν όλες οι πλευρές. Έχουμε ασχοληθεί πολλά χρόνια για το πώς θα μπορέσουμε να προβάλλουμε την ευρωπαϊκή μας διάσταση και την πολιτιστική πολυμορφία στην Ήπειρό μας πώς θα μπορέσει η Ευρώπη του σήμερα να χειριστεί αυτά τα θέματα του πρόσφατου παρελθόντος. Αυτές λοιπόν είναι οι πρωτοβουλίες που θα μας αναγκάσουν να αντιμετωπίσουμε, να αναλύσουμε, να χωνέψουμε και να ε, προχωρήσουμε μπροστά με καλύτερο τρόπο στην Ευρώπη. Η κυρία Κώστα. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Νομίζω ότι αυτή η ιδέα του βραβείου Λουξ ήταν μια πάρα πολύ καλή ε, ιδέα και αυτό αποδεικνύεται σήμερα. Εγώ είδα την ε, ε, Ουγγρική ταινία με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και είμαι βεβαία ότι το ίδιο ενδιαφέρον θα παρουσιάζουν και οι άλλες ταινίες. Νομίζω ότι είναι και μια καλή ευκαιρία για τους βουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου να κατανοήσουν ε, τις ανησυχίες ε, των νέων σκηνοθετών ε, και να ανοίξουν επομένως έναν διαβλό επικοινωνίας που πρέπει να είναι πάντοτε ανοιχτός. Να πω ότι το ε, παράδειγμα που δίνεται εδώ είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον ε, και μπορούμε επομένως να καταρτήσουμε έτσι ένα κατάλογο βέλτιστων πρακτικών ε, στην Ευρώπη. Και πρέπει να σας πω ότι τουλάχιστον εμείς, εγώ από τη δικιά μου πλευρά και στη δικιά μου χώρα θα προσπαθήσω να δημιουργήσω ακόμα ένα κρίκο που θα προσθεθεί στην αλυσίδα αυτή. Νομίζω ότι εδώ ακούσαμε ανθρώπους που έχουν σπρώξει το βλέμμα τους λίγο πιο πέρα από τα σύνορα. Είτε πρόκειται για σύνορα γεωγραφικά, είτε πρόκειται για σύνορα πολιτικά ή ε, κοινωνικά. Ε, και ε, έσπρωξαν λοιπόν το βλέμμα τους πέρα από σύνορα καταδεικνύοντας μια ευαισθησία ιδιαίτερη. Βεβαίως και υπογραμμίστηκε ήδη ότι ήδη και το γεγονός ε, της, ε, του γυρίσματος ταινιών υπερεθνικών ήδη από μόνο του είναι ένα πάρα πολύ μεγάλο ε, πράγμα. Εμείς είμαστε μια επιτροπή που ασχολείται με τον πολιτισμό και επομένως θέλουμε να καταλάβουμε τι πρέπει να κάνουμε παραπάνω στο πεδίο αυτό. Ας πούμε, ε, στην ε, Ιταλία ξέρουμε ότι πρέπει να κάνουμε ένα βήμα όσον αφορά την ψηφιοποίηση των ταινιών και επίσης ε, όσον αφορά την καλύτερη προώθηση και διανομή ταινιών που συνήθως δεν διανέμονται στις μεγάλες αίθουσες. Στην ε, Ρώμη έχουμε και την ε, γιορτή του Διεθνούς ε, Κινηματογράφου και θα ζητήσω στα πλαίσια του φεστιβάλ αυτού να δημιουργηθεί ένα τμήμα που θα αφορά στις ταινίες Λουξ. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε. Είναι μεγάλη τιμή για μας που έχουμε εδώ τόσο μεγάλους σκηνοθέτε και ηθοποιούς. Δεν είδα τις ταινίε, αλλά αύριο θα δω δύο. Δεν θέλω να τις χάσω. Μια που είσαστε εδώ όμως, θα ήθελα, μετά από αυτά που είπε η κυρία Κώστα, και εγώ να κάνω μια ερώτηση. Γιατί βλέπετε στην Ισπανία, τουλάχιστον, είναι δύσκολο να δει κανεί ευρωπαϊκό κινηματογράφο. Για να δει κανεί ευρωπαϊκό κινηματογράφο, μια βουλγαρική ταινία ή δεν ξέρω από ποια άλλη χώρα, είναι πάρα πολύ δύσκολο ως αδύνατο. Είναι κρίμα. Γιατί είναι κάτι που μοιραζόμαστε μεταξύ μας, κάτι που έχουμε κοινό, που δείχνει ακριβώς αυτήν την ε, πολιτισμική πολυμορφία που έχουμε στην Ευρώπη, αλλά δυστυχώς είμαστε υποχρεωμένοι να βλέπουμε συνέχεια αμερικανικές ταινίε. Και νομίζω ότι σε πολλές χώρες ισχύει αυτό, ότι είναι πολύ δύσκολο να δούμε ευρωπαϊκό κινηματογράφο τι θα μπορούσαμε να κάνουμε, τι θα μπορούσε να κάνει η Κομισιόν, το Κοινοβούλιο, ώστε να υπάρχει μεγαλύτερη διανομή, πιο εύκολα διανομή τέτοιων ευρωπαϊκών ταινιών στις χώρες μας. Ο... Η κυρία Χάνιμπολ, ο κύριος Μπίσκι, Χάνιμπολ και μετά ολοκληρώνουμε. Ευχαριστώ. Και εγώ θα ήθελα να καλωσορίσω όλους τους δημιουργούς, τους κινηματογραφικούς δημιουργούς και τους ευχαριστώ ιδιαίτερα που ήρθαν. Αυτή η πρωτοβουλία είναι εξαιρετική και ενθαρρυντική. Ενθαρρύνει τη δημιουργία ευρωπαϊκών ταινιών σε πάνω σε δύσκολα θέματα, πάρα πολύ δύσκολα θέματα. Δεν είναι εύκολο να αντιμετωπίσουμε αυτά τα θέματα τα οποία προβάλλονται μέσω του έργου σας και ε, πιστεύω ότι το επίτευγμά σας είναι σπουδαίο. Όσον αφορά τη διανομή τώρα, ε, ξέρουμε περισσότερα για το ε, τι γίνεται στην υπερατλαντική, από τον, στην υπερατλαντική πλευρά από ό,τι γίνεται στην Βρετανική. Εγώ θα ήθελα να ξέρω πώς θα διανεμηθούν αυτές οι ταινίες. Η διανομή με απασχολεί. Δεδομένου ότι εδώ έχουμε να προσφέρουμε ε, πλούσιο έργο, πρέπει να ξέρουμε πού θα κατευθυνθεί. Ε, πέραν των ε, λίγων εκατοντάδων ευρωβουλευτών και του, των θεατών εδώ μέσα στο σώμα, θα ήθελα να ξέρω πώς θα μπορέσει να, να διαδοθεί αυτή η δημιουργία, αυτά, αυτά τα έργα αλλού, πώς θα διανεμηθούν, τι κανάλια θα ακολουθήσουν, πώς θα αντιμετωπίσουμε αυτή τη διαδικασία διανομής καλύτερα. Ευχαριστώ. Ο κύριος Μπίσκι και μετά πολύ σύντομα ο Χάνο. Η, το βραβείο Λουξ είναι μια εξαιρετική ιδέα και μέχρι τώρα είχαμε μια πάρα πολύ καλή παραγωγή σε ταινίες ε, φοιτητικές υπήρχαν πικρά ε, φεστιβάλ ε, και, και ζει στην πρώην Ανατολική Ευρώπη και είχαμε εξαιρετικές παραγωγές από εκείνη την πλευρά. Ε, ε θα ήθελα συγχαρώ και το Ινστιτούτο Γκιούτε, το οποίο υποστηρίζω ένθερμα, είμαι με, θερμός οπαδός του Ινστιτούτου Γκιούτε. Μέχρι τώρα οι προσπάθειές μας να προβάλλουμε τις ευρωπαϊκές ταινίες δεν ήταν τόσο επιτυχής ε, όσο θα θέλαμε. Έχω παρακολουθήσει τις εξελίξεις τις τελευταίες δεκαετίες. Ε, τι κάνουμε με τις ευρωπαϊκές ταινίες. Δεν χρειαζόμαστε ευρωπαϊκά βραβεία. Δεν χρειαζόμαστε κίνητρα για να μπορέσουν να επιβιώσουν τα μικρά ε, σινεμά τέχνης, τα οποία σιγά σιγά κλείνουν και φθήνουν και εξαφανίζονται. Όχι λοιπόν μόνο ε, χρήματα για παραγωγές, αλλά και χρήματα ε, για τους ανθρώπους που θα προβάλλουν τις ταινίες αυτές. Υπάρχει καμία πρωτοβουλία στήριξης ή ενίσχυσης των κινηματογραφικών αιθουσών, των σινεμάδων δηλαδή όπως λέμε, για να προβάλλουν τις ταινίες αυτές, τις βραβευμένες. Η κυρία Πακ, ε, το κοινοτικό σινεμά, η κοινοτική κινηματογραφική αίθουσα προβολής, το έχουμε ήδη συζητήσει αυτό σαν θέμα. Ο, ο Χάνο τώρα στα φιλανδικά. <laughs> θα χρησιμοποιήσω. Θα μιλήσω στην ε, μητρική μου γλώσσα. Προσέξτε λοιπόν. Πολύ σύντομα. Θέλω να σας πω ότι εκ μέρους της ομάδας μου, των φιλελεύθερων δηλαδή, θέλω να συγχαρώ από βάθος καρδίας όλους τους κινηματογραφιστές που ήρθαν εδώ. Για μένα όλοι έχετε κερδίσει. Συγχαρητήρια λοιπόν. Σας ευχαριστώ που ήρθατε. Νομίζω ότι οι ταινίες οι φετινές είναι πάρα πολύ ενδιαφέρουσες και δίνουν μια πολύ ιδιαίτερη πτυχή όσον αφορά την ευρωπαϊκή διάσταση. Για μένα ο ευρωπαϊκός κινηματογράφος είναι κάτι πολύ σημαντικό. Θέλω να σας ανθαρρύνω να συνεχίσετε τη δουλειά σας και να ξέρετε ότι εδώ στη δικιά μας Κοινοβουλευτική Επιτροπή θέλουμε να προωθήσουμε τον ευρωπαϊκό κινηματογράφο. Το ξέρουμε ότι έχουμε δημιουργούς με ιδιαίτερα προσόντα Μπορεί να έχουμε διαφορετικό κινηματογραφικό λόγο, αλλά αυτό πρέπει να φανεί πολύ περισσότερο από ό,τι γίνεται μέχρι τώρα. Οπότε σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τις προσπαθίες σας. Πολύ σύντομα, ο κύριος Ακίν. Αν θέλετε κάτι να αλλάξετε, εάν το θέλει η καρδιά σας πραγματικά, πρέπει να κάνετε την εισαγωγή μιας ποσόστοσης για ευρωπαϊκές ταινίες. Ποσόστοση Εάν θέλω εγώ στη Γερμανία να δω πορτογαλικά έργα, ισπανικά έργα, ολλανδικά, αλλά δεν μπορώ να τα δω γιατί δεν υπάρχουν αυτές τις ταινίες. Δεν γίνονται, δεν γυρίζονται. Εάν λοιπόν θέλετε να γυρίζονται τέτοιες ταινίες, ε, κάνετε, βάλτε ποσοστώσεις, δώστε ποσοστώσεις. Η Γαλλία το κάνει αυτό με το, το γαλλικό κινηματογράφο. Εάν πάτε σε ένα multiplex σινεμά που, που έχει 12 αίθουσες προβολής θα δείτε ότι και οι 12 παίζουν αμερικανικές ταινίες. Ε, αν δείτε σε, μια ταινία, σε ένα κατάστημα το οποίο πουλάει DVD θα πρέπει να αγοράσετε ταινίες DVD ευρωπαϊκές, ευρωπαϊκές ταινίες σε DVD. Ε, εάν πράγματι θέλετε να επιτύχουμε πρέπει να βάλετε ένα ε, ε, ε, ένα πλαίσιο, να, το ποσοτικοποιήσετε με ποσόστοση το θέμα αυτό και να πείτε χ αριθμός ή ένα χ ποσοστό ταινιών θα είναι ευρωπαϊκές, του ευρωπαϊκού κινηματογράφου. Πάει τελείωσε. Και επίσης θα πρέπει να δώσετε χρήματα σε ένα ευρωπαϊκό ταμείο Έχουμε βεβαίως την χιονοστιβάδα των Αμερικανικών ταινιών, διότι από πίσω υπάρχουν βουνά αμερικανικών ε, πιστώσεων, έτσι, βουνά δολαρίων. Λοιπόν, εάν θέλετε να επιτύχει, θα πρέπει να υπάρχει μία ποσόστοση για τις αίθουσε, μία ποσόστοση διαφημιστικής προβολής και βεβαίως για την παραγωγή, αλλιώς δεν γίνεται. Ευχαριστώ, λέει η Πρόεδρος. Ναι, τι να τα κάνουμε τα χειροκροτήματα. Το Πρόβλημα είναι ότι τόσο γρήγορα και μόνο με ποσοστώσεις δεν μπορούμε να το λύσουμε. Όπου έχουμε κάνει επιβάλλει ποσοστώσεις θα είχαμε αρνητικές αντιδράσεις. Αυτό που μπορούμε να κάνουμε είναι να υποστηρίξουμε το σινεμά της γειτονιάς, να υποστηρίξουμε την καλύτερη διανομή, δεν νομίζω ότι γενικά μπορούμε να κάνουμε εισαγωγή ποσοστώσεων, ποσοτικοποίηση δηλαδή του, της παραγωγής. Ξέρετε ότι όταν προσπαθήσαμε να κάνουμε εισαγωγή ποσοστώσεων και για την εργασία των γυναικών συμμετοχή κλπ, δεν είχαμε και μεγάλη υποστήριξη. Ναι, αλλά η Γαλλία έχει αυτή την ποσόστοση για να ενισχύσει το, το γαλλικό σινεμά. Και έχει επιτύχει καλά, έχει δουλέψει πολύ καλά το σύστημα. Ναι, ναι, αλλά δεν σημαίνει αυτό ότι πρέπει να σπαστούμε οτιδήποτε γαλλικό και αυτό είναι ένα πρόβλημα στην Ευρώπη. Βεβαίω είναι στην Ευρώπη η Γαλλία, δεν λέω. Αλλά δεν νομίζω ότι είναι ο πιο σοφός, ο πιο φρόνιμος τρόπος να προχωρήσουμε. Πρέπει να είμαστε προσεκτικοί, πρέπει να, δούμε πώς μπορούμε να προχωρήσουμε τον ευρωπαϊκό κινηματογράφο και όχι τον εθνικό, όπως η Γαλλία. Ο κύριος Σμιτ. Εγώ συμφωνώ με τον ε, Φατίχ. Το σινεμά τέχνης, οι αίθουσε ε, και το σινεμά τέχνης ε, υποφέρει, έτσι, φθήνει. Στη Γερμανία η κατάσταση είναι πάρα πολύ άσκημη, κλείνουν συνέχεια. Χρειάζεται λοιπόν μεγάλη υποστήριξη για... και, και θέληση και βούληση για να ενισχυθεί το σινεμά τέχνης, ο κινηματογράφος τέχνης και οι αίθουσε με κονδύλια. Ε, ε, θέλουμε, ο στόχος μας είναι να προβάλλουμε σε ευρωπαϊκές χώρες ευρωπαϊκές ταινίες και εν συνεχεία προχωρήσουμε και πιο έξω. Σωστό, λέει η Πρόεδρος. Ε, πολύ μεγάλο θέμα. Θα το συζητήσουμε ξανά. Πιστεύω ότι έχουμε μία βάση συζήτησης. Η σύμβαση της UNESCO είναι ακριβώς ένα μέσο το οποίο μας δίνει αυτά τη δυνατότητα και πρέπει να το σκεφτούμε αυτό. Ε, θα κάνουμε μία ακρόση σύντομα ε, για το θέμα των ε, ρητρών εξαίρεσης και των εξαιρετικών ρυθμίσεων μέσω της UNESCO και σας υπόσχομαι ότι θα φέρουμε το θέμα αυτό στην ημερήσια διάταξη. Μόνο που δεν μπορώ να σας υποσχεθώ τι αποτέλεσμα θα έχουμε. Εκεί που μπορέσαμε κάτι να κάνουμε είναι ακριβώς το βραβείο Lux και γι' αυτό ακριβώς έχουμε ε, οργανώσουμε αυτή τη συνάντηση. Σημειώσαμε τα αιτήματά σας. Έχουμε καιρό, μήνες και χρόνια, πέντε χρόνια είναι η σύντια μας, να προχωρήσουμε και να ε, ενισχύσουμε τη διάσταση αυτή του Ευρωπαϊκού Κινηματογράφου. Θα ήθελα τώρα να ολοκληρώσω αυτή τη συνεδρίαση. Σας ευχαριστώ όλους τους καλεσμένους μας που ήταν και μας τίμησαν. Με την, παρουσία, με την παρουσία τους Τονίζω ξανά ότι αυτή ήταν μια εξαιρετική